Right, welcome. Καλώς ορίσατε. Παρακαλώ καθίστε. Okay, thank you very much. Σας ευχαριστώ πολύ. ανακοινώνω την ε, εκκίνηση αυτή της ε, συνεδρίαση. Πρώτα απ' όλα τα ε, έγκριση της ημερήσιας διάταξη Υπάρχουν αντιρρήσεις, όχι. Η ημερήσια διάταξη λοιπόν έχει εγκριθεί με τις ανακοινώσεις της Προέδρου για την ακρόαση για το MIFID. Ζητώ συγγνώμη από τους ομιλητές για το γεγονός ότι δεν θα προεδρεύσω την ίδια την ακρόαση Μόλις επέστρεψα από τις Ηνωμένε Πολιτείε, όπου παρέστην στο Διατλαντικό Διάλογο Νομοθετών, όπου συζητήθηκα μεταξύ άλλων και οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με τους νομοθέτες των ΗΠΑ. Αρκετά σημαντικό το θέμα. Θα αναθέσω λοιπόν στην ε, κυρία Μακάρθη την ακρόαση καθώς αυτή είναι η συγγήτρια για την οδηγία κατάχρησης των αγορών και για το ε, MIFID από την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς. Την ενδιαφέρει λοιπόν ιδιαίτερα αυτός ο φάκελος. Επίσημα θα πρέπει να σας αναφέρω για τον τριμερή διάλογο. Ο πρώτος έλαβε χώρα στις 28 Νοεμβρίου κάλυψε πολλά ζητήματα και επετεύχθη κάποια πρόεδρος. Ο επόμενος τριμερής διάλογος θα λάβει χώρο στο Στρασβούργο την εβδομάδα της 12ης Δεκεμβρίου. Δεν έχει οριστεί ακόμη χρονική στιγμή. Το σύστημα διασφαλίσεων για καταθέσεις, ο, τριμερής διαλόγος έλαβε χώρα και έγινε η πρώτη συνεδρίαση σε τεχνικό επίπεδο την 1η Δεκεμβρίου. Είχε να κάνει με μη πολιτικά θέματα. Σημειώθηκε ικανοποιητική πρόοδος και στις δύο συνεδριάσεις και ένας ενημερωμένος πίνακας θα διατεθεί στις πολιτικές ομάδες εν ευθέτω χρόνο η επόμενη τριμερής συνεδρίαση θα λάβει χώρα στις 13 Δεκεμβρίου στο Στρασβούργο. Όσον αφορά το ΣΕΠΕΡ, ένας τέταρτος ε, διάλογος έλαβε χώρα στις 13 Νοεμβρίου με μια προσωρινή συμφωνία όπου και η Κομισιόν και το Συμβούλιο συμφώνησαν να επανεξετάσουν η συμφωνία αυτή αφορούσε στη χορήγηση στα κράτη-μέλη μιας παρέτησης για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και ε, μια ημερομήρια πιο νωρίς ε, όσον αφορά τη διακυβέρνηση και τα δικαιώματα ε, αποζημίωσης. Το Συμβούλιο μπορεί να συμφωνήσει. Το κείμενο έχει διευθετηθεί, έχει συμφωνηθεί. Όσον αφορά τις δηλώσεις που αποτελούν ουσιώδες κομμάτι για το Κοινοβούλιο, οι ενδείξεις ε, προς το παρόν είναι λιγότερο ενθαρρυντικές Εφόσον επιληθεί το ζήτημα με τις δηλώσεις, στις 15 Δεκεμβρίου θα μπορέσει να συμφωνηθεί το κείμενο και θα ξανασυμβολευτούμε αυτή την Επιτροπή βάσει κανόνα 73 στις 19 Δεκεμβρίου με στόχο την Ολομέλεια του Φεβρουαρίου. Αυτή τη στιγμή λοιπόν αναμένουμε την πλήρη συμφωνία με την Κομισιόν. Σας ζητώ συγγνώμη τώρα λοιπόν που χρειάζεται να αναχωρήσω. Θα παρακολουθήσω το web stream ε, με την ησυχία μου μια άλλη μέρα και δίνω τον λόγο ε, και τη θέση του Προέδρου στον κύριο Μακάρθη. Ευχαριστώ. Στην κυρία Μακάρθη. Uh, well, colleagues, because my, my voice αγαπητοί συνάδελφοι. Επειδή έχει κλείσει λίγο η φωνή μου, δεν θα μιλήσω πολύ. Χωρίς καθυστέρηση λοιπόν. Πιστεύω καταλαβαίνετε από το πρόγραμμα. Έχετε δει πως έχει χωριστεί σε τρεις ενότητες η ακρόαση. Έχουμε κάποιους ε, πολύ καλούς εμπειρογνώμονες μαζί μας σήμερα. Πρώτα απ' όλα ήθελα να δώσω λόγο στον εισηγητή μας, τον κύριο Φέρμπερ ώστε να μας κάνει τις αρχικές παρατηρήσεις και τα σχόλιά του. Ευχαριστώ Πρόεδρε και αγαπητοί συνάδελφοι. Καλημέρα σας. Χαίρομαι ιδιαίτερος που μπόρεσαν να έρθουν κάποιοι λίγοι συνάδελφοι. Βλέπουμε γενικά άδεια έδρανα στο κέντρο της αιθούς, αλλά εν πάση περιπτώσει ελπίζω ότι θα έχουμε αρκετή προσοχή εξασφαλίσει. Αποτελεί ένα επίκεντρο, μια, μια αφετηρία για την επεξεργασία μια νέα οδηγία ύστερα από τις προτάσει Ευρωπαϊκή Επιτροπής ε, ε, στι αρχέ Οκτωβρίου αυτή η συνεδρίαση και η Επιτροπή μας πιστεύω τους τελευταίους μήνες έχει καταλήξει μια σειρά από μέτρα, φερρυπίν, ε, εποπτικές αρχές, εποπτική αρχή για τις τράπεζες, για τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, χρεογράφων και νομοθετήματα όπως σε παραδείγματι εναλλακτικά επενδυτικά κεφάλαια για τα παράγωγα over the counter, ελευθερής ε, πώληση δηλαδή και το καθεξής. Ωστόσο, μπορούμε να πούμε ότι προχωρούμε σε ένα ακόμη πολύ σημαντικό κομμάτι για τη ρύθμιση των αγορών, διότι έτσι μπορούμε να εξασφαλίσουμε πολύ σημαντική διαφάνεια, προστασία του καταναλωτή και ισότιμες συνθήκες ανταγωνισμού στις χρονοπιστωτικές αγορές. Ως ηγητής, εγώ θεωρώ πολύ σημαντικό το να υπάρξει διαφανής μέθοδος εργασίας στην επεξεργασία του θέματος αυτού, το οποίο κρίνω τόσο σημαντικό. Και γι' αυτό είναι καλό να ξεκινήσουμε με αυτή την ακρόαση, όπου μπορούμε να ανταλλάξουμε απόψεις με διαφόρους ειδικού σε διάφορους τομείς, για να συλλέξουμε τις πληροφορίες από πλευράς τους. Έχω μιλήσει και με τους κοιόδης ηγητές από τις άλλες ομάδες και έχουμε ε, καταρτήσει ένα ερωτηματολόγιο το οποίο έχει δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της Επιτροπής μας και το οποίο έχουμε αφήσει μέχρι τις 13 Ιανουαρίου ανεκτό, δηλαδή δίνουμε τη διπλάσια, ε, το διπλάσιο περιθώριο διαβούλευσης από αυτό που προσέφερε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μέσα σε αυτό μπορεί να κάνει κανείς παρατηρήσεις του, όπως είπα, μέχρι τις 13 Ιανουαρίου. Αυτή θα είναι η διαδικασία συναπόφασης ή διαβουλεύσεων καλύτερα του Κοινοβουλίου και έτσι μπορούμε να έχουμε στο δυνατόν πιο διαφανεί διαδικασίες. Σήμερα έχουμε καταθέσει ένα πρώτο έγγραφο εργασία. το βλέπετε στους φακέλους σας φαντάζομαι, το οποίο αποτελεί μια συμπίληση των ε, προτάσεων που έχουμε ήδη, των, ε, ισχυουσών, των ισιών, των νομοθετικών κειμένων και των υπεραιτέρω προτάσεων που πιστεύουμε θα μας επιτρέψουν να συζητήσουμε ε, εστιασμένα τους διάφορους τομείς που μας ενδιαφέρουν για να καταλήξουμε όπως ελπίζω σε μια καλή και ε, ισορροπημένη έκθεση. Στην προετοιμασία της σημερινής συνεδρίασης ε, επικεντρωθήκαμε σε τρεις, βασικούς θεματικούς, σε τρεις βασικές θεματικές ομάδες. Δεν θα επισελθώ σε λεπτομέρειες, άλλωστε υπάρχουν και στο, στην ημερήσια διάταξη. Βέβαια, πάντα σε κάθε τομέα υπάρχει ένας ειδικό, ε, ένας που θα μπορούσε να θεωρηθεί κατάλληλη προσωπικότητα για να μιλήσει στο, στα θέματα αυτά. Ε, θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε πάνω σε καμιά πενηνταριά ονόματα ειδικών, πλην όμως θεώρησα ότι καλό θα ήταν να έχουμε επαρκές περιθώριο για ανταλλαγή απόψεων και γι' αυτό προτίμησα να μην δοθεί ο λόγος στον κάθε έναν ειδικό στο θέμα αυτό, αλλά να δώσουμε τη δυνατότητα μέσω του ερωτηματολογίου που προανέφερα σε όποιον ενδιαφέρεται να συμβάλλει σε αυτή τη διαφανή διαδικασία ε, για τη λήψη της απόφασης των αποφάσεων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και πριν ακόμη από τις προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής είχε μέσα από ένα ψήφισμα τοποθετηθεί στο θέμα αυτό. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Σουίμπλορν, η οποία ο συντάκτρια του ψηφίσματο εκπροσώπησε εδώ και διατύπωσε τι θέσει του Κοινοβουλίου. Πιστεύω ότι μπορούμε να πούμε κατ' ουσίαν ότι βρίσκουμε ικανοποιητικό το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δέχεται μια σειρά από τις προτάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τις προδιαγραφές διαφάνειας, το θέμα το σχετικό με τη συχνότητα των συναλλαγών, όλα αυτά τα οποία θα συστήσουμε φυσικά. Υπάρχουν και πολλά άλλα θέματα στα οποία θα θέλαμε περισσότερη πρόοδο. Από την άλλη υπάρχουν κάποια σημεία τα οποία έχουμε εμείς προτείνει και τα οποία δεν έχει λάβει υπόψη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Φερρυπίν, δεν προβλέπεται νέος ορισμός αγοράς για τις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές. Πράγμα δεν ζητούσε το Κοινοβούλιο δηλαδή ειδικό ορισμό, πράγμα το οποίο όμως έπραξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και βέβαια θα πρέπει να δούμε γιατί αυτή η οδηγία πρέπει να προχωρήσει σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Είναι γνωστό πιστεύω της ε, Πάσιν ότι έχει αλλάξει σημαντικά το πεδίο μας στο οποίο δραστηριοποιούνται οι αγορές το τελευταίο, στο τελευταίο διάστημα, τα τελευταία χρόνια και για λόγους τεχνολογικής εξέλιξης αλλά και για λόγους νομοθετικούς. Και έτσι στη συμφωνία του Pittsburgh, τον, του G20 νομίζω ότι συμφωνήθηκε να προχωρήσουμε με αγορές ρυθμισμένες και προϊόντα που, που θα ακολουθούν κάποιους κανόνες. Αυτό νομίζω θα πρέπει να είναι το αντικείμενο των προσπαθειών μας. Οι προτάσεις λοιπόν τις οποίες έχουμε τώρα να συζητήσουμε και να επεξεργαστούμε είναι οι δομές ίδιες της αγοράς ή των αγορών, Υπάρχουν ειδικέ προδιαγραφέ για τι ε, μικρέ και μεσαίες επιχειρήσει, το ζήτημα το οποίο έχει να κάνει με τι αγορέ αγαθών, που επίση θα μα απασχολήσει, στη συζήτηση και όπου πιστεύω έχουμε σημαντικό μερίδιο ε, αρμοδιοτήτων ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Από την εμπειρία άλλωστε που έχουμε και από τα τελευταία χρόνια είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το ζήτημα της ε, ΕΣΜΑ που ασφαλώς θα πρέπει να αναφερθεί επίσης διότι η τεχνική προσαρμογή για την πρώτη οδηγία όπνη που έχει ήδη ξεκινήσει και υπάρχουν ε, και πολλές διατάξεις θα πρέπει να ληφθούν υπόψη, πολλές επιλογές που θα πρέπει να υλοποιηθούν. 35 διαφορετικές συγκεκριμένα είτε εποπτικές είτε εφαρμοστικέ ε, προδιαγραφές σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ένα δείκτη που αποδεικνύει που θα πρέπει να συστήσουμε πολύ επακριβώ το ρόλο τη ΕΣΜΑ και το ενδεχόμενο απαγόρευση προϊόντων, ε, συναλλαγή δηλαδή σε προϊόντα που προτείνεται σχέση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι κάτι το οποίο πρέπει να συζητήσουμε. Το ζήτημα του πεδίου εφαρμογή επίση, ενδεχόμενων παρεκκλήσεων ή εξαιρέσεων, προστασία του επενδυτή από δράσει ε, των, συμβόλων, των συμβούλων επενδύσεων, ε, συναλλαγές υψηλή συχνότητα ή άλλα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις τεχνολογικές εξελίξεις που δεν μπορούν ενδεχομένω να προβλεφθούν ακόμη. Έχουμε να κάνουμε επίση με ρυθμίσεις σχετικές με τρίτο κράτος ή με τρίτα κράτη, με κυρώσεις και άλλα πολλά που δεν θέλω να εκθέσω αναλυτικά. Όλα αυτά δηλαδή τα οποία έχουν να κάνουν με το επίκεντρο ακριβώς των ρυθμίσεων των χρηματοπιστωτικών αγορών και γι' αυτό ευχαριστώ ιδιαίτερως τους συναδέλφους που ε, μας αφιερώνουν το χρόνο του σήμερα αλλά πάνω απ' όλα όσους ήρθαν να μας μιλήσουν στη, στα τρία αυτά, στους αυτούς γύρους της συζήτησης που έχουμε προβλέψει και μπορούμε πιστεύω εφόσον μπορέσουμε να μιλήσουμε για μη fit και μη fear, να προσδιορίσουμε, να καταθέσουμε ένα πρώτο ορόσημο στην πορεία αυτού του νέου νομοθετήματος. Έχουμε ξεκινήσει με τους συναδέλφους ε, τη δουλειά αυτή και τη συνεργασία σε πολύ καλό πνεύμα και πιστεύω ότι και μετά τα Χριστούγεννα θα συνεχιστεί αυτή η αγαστή συνεργασία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Φέρπερ. Έχουμε εδώ όλους τους σκιώδεις. Καλό αυτό. Έχουμε όλους τους ειδικού που είναι έτοιμοι να υποβάλουν ερωτήσεις στους εμπειρογνώμονες μας που έχουμε καλέσει σήμερα εδώ. Ξεκινάμε με το πρώτο τμήμα που είναι το ερώτημα έχουμε τους σωστούς θεσμούς, υπηρεσίες, δραστηριότητες, πλατφόρμες διαπραγμάτευσης και μέσα Πέντε λεπτά θα έχει ο κάθε μιλητή. Σα παρακαλώ να τηρήσετε το χρόνο σα, γιατί αλλιώ θα δυσκολευτούμε να ακούσουμε όλου και να έχουμε και ερωτήσει και απαντήσει. Ο πρώτο είναι ο Κάρε Καρελάνο, που είναι εκλεκτικό διευθυντή του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πολιτικών Μελετών. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ πολύ όλου του ευρωβουλευτέ μέλη τη επιτροπή τη οικονομική που μου δίνετε την ευκαιρία να έρθω εδώ και να σα μιλήσω. Είναι πολύ σημαντικό, όπως είπε και ο κύριος ε, Φέρμπερ, ε, να μιλήσουμε για την οδηγία αυτή. Πάνε τέσσερα χρόνια που έχει ξεκινήσει η οδηγία αυτή και είναι καλό να ρωτιέται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τι έκανε, τι ήθελε μάλλον να πετύχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όταν ε, υιοθετήθηκε η οδηγία αυτή και τι έχει γίνει σήμερα. Έχουν επιτευχθεί οι στόχοι. Έχουν πραγματοποιηθεί στο μεταξύ. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λοιπόν είναι καλό να καταλάβει περί τίνος πρόκειται. Ποια είναι αυτή η αναθεώρηση της οδηγίας MIFID στην αρχή η οδηγία ονομαζόταν Οδηγία για τι Επενδυτικέ Υπηρεσίε. Ίσως ήταν πιο ξεκάθαρο όρο όρος αυτός. Πρόκειτο για κάθε επενδυτική υπηρεσία, για τι διαπραγματεύσει δηλαδή, στις πλατφόρμες διαπραγμάτευση όπω λέγονται, πρόκειται για του ενδιάμεσου τους μεσολαβητές και πρόκειται και για την προστασία του επενδυτή. Αυτά τα τρία ήταν τα βασικά στοιχεία. Τώρα ε, αντικαθίσταται η οδηγία αυτή του 93 που έζησε 10 χρόνια περίπου, μέχρι το 2004 που υιοθετήθηκε η οδηγία Μύφη, αλλά άρχισε να εφαρμόζεται το 2007. Η αρχική οδηγία των ε, επενδυτικών ε, υπηρεσιών είχε ήδη φροντίσει για διάφορες προδιαγραφές, ε, αυτό που δεν έκανε όμω ήταν ότι δεν καταργούσε το μονοπόλιο των εθνικών χρηματιστηρίων. Αυτό γίνεται με την νέα οδηγία, με την μύφη τώρα την οδηγία δηλαδή για τι αγορέ χρηματοπιστωτικών μέσων, που καταργεί τα μονοπόλια αυτά και εισαγάγει δύο νέε κατηγορίε πλατφόρμα διαπραγμάτευση. Η μία είναι ο πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευση και ο δεύτερο είναι ο συστηματικός, η συστηματική μάλλον ιστορικοποίηση. Και έτσι αυτή είναι η βασική αλλαγή που έχουμε σε σχέση με την προηγούμενη οδηγία. Επίση. αυτό όμω που δεν έγινε είναι ότι δεν, ε, το θέμα της διαφάνειας τιμών δεν επεκτάθηκε και στα ομόλογα και στις, ε, στα παράγωγα. Τώρα, πολλά πράγματα δεν εφαρμόζονται πλήρως. Ορισμένες χώρες έχουν πάρει βέβαια κάποια βήματα προς σωστή κατεύθυνση, να συμπεριλάβουν δηλαδή και τα ομόλογα ή τι αγορέ παραγόγων, αλλά όχι όλε. Είμαστε τέσσερα χρόνια λοιπόν μετά τη θέση σε ισχύ τον Νοέμβριο του 2007 της οδηγίας MIFID, η οποία μιλάει για διαπραγμάτευση σε διάφορους τόπους διαπραγμάτευσης. Ε, έχει μειωθεί μεν το κόστος, αλλά δεν έχει καθόλου πληγή η ρευστότητα. Ο εισηγητής το είπε και πριν από λίγο, ότι Έχουμε χρησιμοποιήσει νέες τεχνολογίες προκειμένου να υπάρξει επέκταση στις πλατφόρμες διαπραγματεύσεων και να υποφεληθούμε έτσι από τον ανταγωνισμό. Οι υπάρχουσες διαπραγματεύσεις όντως ε, έχουν ενισχύσει τον ανταγωνισμό, αλλά σε ένα μικρό βαθμό, δεδομένου ότι από τους νέους που έχουν εισαχθεί στο σύστημα, μόνο GX έχει καταφέρει να πάρει ένα σημαντικό μέρος της αγοράς ε, μετοχών και είχαν 30% στα τέλη του Αυγούστου. Το πρόβλημα τώρα παραμένει ότι υπάρχουν πολλές εξαιρέσεις, πολλές απαλλαγές, ότι υπάρχουν ε, πολλοί καινούργοι τόποι διαπραγματεύσεων, κάτι το οποίο οδήγησε και σε χρηματιστηριακά δίκτυα. Τώρα, για την προστασία του επενδυτή, πιστεύω ότι οι επιπτώσεις της οδηγίας δεν είναι τόσο σημαντικές. Ή ας πούμε, ότι η οδηγία όταν άρχισε να ισχύει τον Εύρο το 2007 ε, φαινόταν να ήταν καλά προσαρμοσμένη στις ανάγκες που είχαμε τότε με την εμφάνιση της οικονομικής κρίσης. Τώρα, λίγα χρόνια μετά, μπορούμε να πούμε ότι το στοιχείο κλειδί είναι η βέλτιστη εκτέλεση, η καταλληλότητα του επενδυτή και τα συγκρόμενα συμφέροντα. Πράγματα τα οποία έχουν σχεδιαστεί πολύ καλά μεν, αλλά δεν έχουν εφαρμοστεί ικανοποιητικά. Αυτή είναι μια αποτυχία. Παραμένουν αμφισημίες και έτσι δεν έχουν αντιμετωπιστεί όλα τα θέματα που έχουν να κάνουν με την εφαρμογή της νέας αυτής οδηγίας. Στο μεταξύ βέβαια δημιουργήθηκε η Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή, κάτι το οποίο βοήθησε και άλλα θέματα ε, καλύπτονται από την τροποποίηση της οδηγίας MIFID. Πέρα τώρα από την ε, έρευνα που έγινε, μπορούμε να πούμε και από τα αποτελέσματά της δημοσιεύθηκαν στις αρχές του 2011, φαίνεται ότι τα βασικά θέματα που πρέπει να λυθούν με την εφαρμογή της οδηγίας είναι το θέμα της ποιότητας των δεδομένων και της ε, ενοποίησης και της εφαρμογής των ε, κανόνων θεοντολογίας των επενδυτικών επιχειρήσεων. Η επαλήθευση πάντως της εφαρμογής της βέλτιστης εκτέλεσης είναι κάτι το οποίο παραμένει ως πρόβλημα. Ένα άλλο θέμα είναι το ότι η οδηγία MIFID είναι πολύ καλή. Υπάρχουν οι κανόνες για τα οικονομικά κίνητρα, για τη σύγκρουση συμφερόντων, αλλά παρόλα αυτά δεν έχουν εφαρμοστεί. Οι κανόνες υπάρχουν αλλά δεν εφαρμόζονται. Γι' αυτό η MIFID 2 τώρα έχει προδιαγραφές οι οποίες ενισχύουν τους κανόνες αυτούς. Αλλά παραμένει το θέμα το κατά πόσο θα εφαρμοστούν υπάρχοντες κανόνες. Η πιο σημαντική αποστολή πάντως της MIFID 1 ήταν ε, το θέμα της ε, διαφάνειας στις ε, διατάξεις και στην εφαρμογή των διαπραγματεύσεων τίτλων. Η επέκταση στα ομόλογα είναι κάτι το οποίο συζητήθηκε. Νομίζω τώρα ότι έπρεπε να έχει γίνει. Ήταν κρίμα που δεν έγινε και ελπίζω τώρα η διαφάνεια αυτή τη τιμών να επεκταθεί και στην αγορά την έξω χρηματιστηριακή παραγόγων. Η Μίφιτ έπρεπε ήδη να το είχε προβλέψει. Τώρα το προτείνει πάντως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να υπάρξουν και οι υπηρεσίες διακανονισμού δηλαδή για τα CDS. Τώρα πάμε πίσω το 2007 η ΜΥΘΙΤ φαινόταν ότι θα έλυνε ε, το θέμα της εξέλιξης στην ε, αγορά την ευρωπαϊκή. Αλλά ο καιρός περνάει γρήγορα. Οι εταιρείε αρχίζουν τώρα να βλέπουν ότι πρόκειται για μια νέα ευκαιρία. Η οδηγία όντως ενίσχυσε την αποτελεσματικότητα και τον ανταγωνισμό στις ευρωπαϊκές οικονομικές αγορές και αντιμετωπίζει βοηθάει να αντιμετωπιστούν και τα πρόβλημα από την οικονομική κρίση. Νομίζω ότι πρέπει να παραμείνει και να φροντίσει να μην υπάρξουν υπερβολικά πολλές ρυθμίσεις στους χώρους διαπραγμάτευσης τίτλων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ζητήσω τον κύριο Φιλιππονάκης, ε, ε, Finance Watch. Ευχαριστώ πολύ. Για να απαντήσουμε το ερώτημα σήμερα θα έχω στο νου μου τους στόχους της MIFID για την καθιέρωση ενός πιο ασφαλούς, πιο υγιούς, πιο διαφάνους ε, συστήματος χρηματοοικονομικού που θα εξυπηρετεί την οικονομία και την κοινωνία στο σύνολό τη. Εξετάζοντας το κατά πόσο η MIFID έχει επιτύχει ε, να, το στόχο της ικανοποίησης ε, της ζήτησης ε, από τα συστήματα, τα χρηματοοικονομικά με τρία κριτήρια. Το ένα είναι διαφτερό με την καλύτερη δυνατή τιμή και τρίτη με στόχο επικεντρωμένη στην εξυπηρέτηση της πραγματικής οικονομίας και της κοινωνίας. Ας δούμε πρώτα την διαφάνεια. Πρώτα απ' όλα τα δεδομένα. Περίπου 40% των μετοχών σήμερα ε, αποτελούν το αντικείμενο εξοχρηματιστηριακής διαπραγμάτευσης συν 6% ε, των μετοχών από τα dark pools. Αυτό σημαίνει ότι το 46% της αγοράς μετοχών στην Ευρώπη ε, αποτελούν το αντικείμενο διαπραγμάτευσης χωρίς πληροφορίες πριν από τη διαπραγμάτευση. Πέρυσι λάβαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα εκθέση από το Πανεπιστήμιο της Φραγκφούρτης όπου αναφερόταν ότι 39% όλου των διαπραγματεύσεων OTC για μετοχές βρίσκονταν κάτω από το μέγεθος που προέβλεπε η MIFID. 9% είναι, έχουν το τυπικό μέγεθος ε, της αγοράς ε, το οποίο σημαίνει ότι αν προσθέσουμε το 39 με το 9, 48% των εξωχρηματιστηριακών διαπραγματεύσεων είναι κάτω από το ε, στάνταρ ε, μέγεθος της αγοράς. Θα σας υπονθυμίζω ότι μεγάλο μέγεθος είναι το μέγεθος που αφορά αυτό που ονομάζουμε dark pool trading ε, όπου υπάρχει λιγότερη διαφάνεια άλλο ένα 39% των OTC είναι μεγαλύτερου μεγέθους. Το 37% των συναλλαγών OTC παραβιάζουν ουσιαστικά το πνεύμα της MIFID. Όχι τις προδιαγραφές. Οι προδιαγραφές δεν ήταν ιδιαίτερα ισχυρές ε, ε, τότε. Δεν είναι δηλαδή παράνομες, αλλά παραβιάζουν το πνεύμα της διαφάνειας των ελεύθερων συναλλαγών που αποτελούσε την ουσία της MIFID 1. Συνεπώς οι ανησυχίες μας για τη μη διαφανή αγορά υπάρχουν ακόμα, ισχύουν ακόμα και σίγουρα η οικονομική ωφέλεια δεν πρόκειται να βελτιωθεί αν δεν διορθώσουμε αυτή την κατάσταση. Το δεύτερο κριτήριο είναι η καλύτερη δυνατή τιμή. Όπως αναφέρει ο προκάτοχος της ΕΣΜΑ το 2009 έλεγε ότι ο κατακριματισμό της αγοράς έχει οδηγήσει σε μεγαλύτερο αριθμό εκτελέσεων σε πολλούς τόπους που αυξάνει τελικά το κόστος των συναλλαγών. Ουσιαστικά το κόστος των συναλλαγών έχει αυξηθεί, το κόστος των συναλλαγών έχει μειωθεί, αλλά ουσιαστικά η τιμή που πληρώνουν οι επενδυτές είναι υψηλότερη. Τα στατιστικά στοιχεία είναι λίγο παλιά έχουν γίνει προσπάθειες ενημέρωσης, αλλά θα πρέπει να αναρωτηθούμε κατά πόσο τα στατιστικά στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας είναι, ακόμη ισχύουν. Περνάω στο τρίτο σημείο, το κατά πόσο εξυπηρετούμε καλύτερα την οικονομία και την κοινωνία. Γνωρίζουμε ότι ο κατακαιρματισμός της αγοράς έχει βοηθήσει στην ανάπτυξη της, ε, των συναλλαγών υψηλή συχνότητα σε ποσοστό 35% των συναλλαγών επιμετοχών στην Ευρώπη. Η HFT είναι ένα αποσύνολο της των αλγοριθμικών συνολογών. Πρόκειται για διατησία τιμών μεταξύ διαφόρων τόπων. Υπάρχουν επίσης στρατηγικές που βασίζονται σε διαφορετικές πρόσβασεις, σε πληροφορίες για τις τιμές και σε μερικές περιπτώσεις μιλάμε και για κατάχρηση της αγοράς. Όχι πάντα φυσικά, αλλά ορισμένες φορές ε, έχουμε ε, παραπλάνηση διάφορες τεχνικές. Πρέπει να γίνει διάκριση. Είναι πολύ σημαντικό μεταξύ HFT που δημιουργούν ρευστότητα και HFT που δημιουργούν όγκο. Υψηλή συχνότητα δηλαδή συναλλαγές που δημιουργούν ρευστότητα και που δημιουργούν όγκο. μόνο η HFT που σχετίζεται με ε, τις αγορές δημιουργεί ρευστότητα, ενώ όλες οι άλλες μορφές ε, δημιουργούν όγκο, όπως συνέβη στην περίπτωση του Flash Crash της ΕΠΑ το 2010, όπου συμβάσεις ε, μετοχών ε, αξίας 7, εκατομμυρίων, 7 δισεκατομμυρίων δολαρίων άλλαξαν χέρια 27.000 φορές σε 14 δευτερόλεπτα με αποτέλεσμα την κατάρρευση της αγοράς. Αυτό έδειξε ότι το μέγεθος των συναλλαγών HFT ενισχύει προϋπάρχουσες ε, τάσεις και καθοδηγεί το ενδιαφέρον των επενδυτών. Εμείς έχουμε συζητήσει πολλές φορές ε, τους ε, τελικούς επενδυτές και έχουμε αποδεικτικά στοιχεία όπου τελικοί επενδυτές μας λένε ότι πολλές φορές τους, τους ξεπερνούν οι HFT όσον αφορά τις αναλλαγές. Οι συναλλαγέ υψηλή συχνότητα. Θα πρέπει να κάνουμε διάκριση των συναλλαγών υψηλή συχνότητα που φέρνουν ρευστότητα και των ε, HFT που ε, δημιουργούν όγκο. Ω συμπέρασμα, παρά τι προθέσει τη η ΜΕΦΙΝΤΑΒ 1 δεν έχει βελτιώσει τη δικαιοσύνη, τη διαφάνεια, τη ρευστότητα και την ανταγωνιστικότητα τιμών στην αγορά με αποτέλεσμα τη βελτίωση της προστασίας των ε, επενδυτών. Έχουν γίνει κάποια βήματα προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά απέχουμε ακόμη πολύ. Πιστεύουμε τελικά ότι η έκθεση που ενέκρινε τον Εύρο του 2010 ε, η Σχετική Επιτροπή περιλαμβάνει χρήσιμες προτάσεις που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στη διαδικασία MIFID. Εμείς στη Finance Watch θα υποβάλουμε συγκεκριμένες προτάσεις για το θέμα που αναφέραμε σήμερα και άλλα θέματα που δεν εξετάζουμε όπως την προστασία των επενδυτών και τις υπευθύνες πωλήσει. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό τον αρκτήριο λάκτισμα. Κρατάμε και το χρόνο μας. Κύριε Φέρμπερ, έχετε κάποιες ερωτήσεις για να ακούσουμε μετά τους σκιώδεις. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δύο πράγματα μόνο, έχει πολλές ερωτήσεις. Πρώτον, στην πρόταση της Επιτροπής υπολογίζεται στο, χώρο, στο πεδίο εφαρμογή και το πιστοποιητικό εκπομπών. Θα ήθελα λοιπόν αυτό να το διευκρινίσουμε και για τον κύριο Φίλιππο Νάζη για το εμπόριο της συναλλαγής υψηλής συχνότητας. Θα πρέπει να δούμε αφενός με τη ρευστότητα αφετέρου δε την ε, χρήση των αλγορίθμων και την ευστάθειά τους. Ε, και θα ήθελα να πω ότι μερικές φορές δεν είναι πολύ σαφή όλα αυτά τα πράγματα ως συμπέρασμα δηλαδή αυτό που έχει καταγράψει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιστεύετε ότι είναι ικανοποιητική απάντηση για την αποφυγή ενός ενδεχόμενου flash crash ή πιστεύετε ότι δεν επαρκεί αυτές οι δύο σύντομες ερωτήσεις μόνο για μένα ευχαριστώ Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρο. Κύριε Φέρμπερ, αν δεν έχετε αντίρρηση, θα έλεγα αντί να κάνουμε ερώτηση και απόκριση, να Κάνουμε ένα γύρο ερωτήσεων και μετά εσείς τι πρόεδρος, πρόεδρο, τι θέλετε. Βεβαίως, όχι, για να έχουμε δώσει το δυνατόν καλύτερη, να αξιοποιήσουμε καλύτερα το χρόνο αυτής της ακρόασης. Κύριε Γκέβελς, παρακαλώ εσείς τότε. Ναι, ευχαριστώ πρόεδρε. Δύο στόμες ερωτήσεις μόνο. Για τη διαφάνεια, καταρχάς. βλέπω εκπροσώπους διαφόρων ομάδων επενδυτών που πάντα λένε ναι βεβαίως διαφάνεια αλλά όταν ε, προσπαθούμε να ελέγξουμε τις συναλλαγές τύπου τις, τις ελεύθερες συναλλαγές δηλαδή αυτές που δεν υφίσταται κανένα έλεγχο που δεν έχουν παρουσιάζουν δηλαδή διαφάνεια και η Ευρωπαϊκή, Επιτροπή προσπαθεί να προτείνει τα OTF ερωτώ, αυτά τα OTF μπορούν να αποτελέσουν αντίδραση στο over the counter. Μπορούν να δώσουν τη λύση και τη διαφάνεια σε αυτές τις συναλλαγές. Δεύτερο, συχνότητα, συναλλαγές υψηλής συχνότητας. Εγώ θεωρώ ότι οι αγορές ιδρύθηκαν, ε, στάθηκαν και υπάρχουν για να επιτρέπουν στον συναλλασσόμενο να αναζητά την ε, τιμή που τον ενδιαφέρει. Αλλά αυτό πού μπορεί, πώς μπορεί να υφίσταται να λειτουργεί εάν μέσα σε δευτερόλεπτα μπορεί ένας ε, ηλεκτρονικός υπολογιστής να καταγράψει αλλαγές ε, σε τιμές χωρίς κανείς να έχει τη δυνατότητα να ε, ελέγξει ή να παρακολουθήσει αυτές τις εξελίξεις στις τιμές. Έτσι λοιπόν ε, αυτές οι ε, υψηλή συχνότητα συναλλαγέ δεν θα έπρεπε να υπαχθούν κατά κάποιο τρόπο σε αλγοριθμικέ συναλλαγέ. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρο. Ε, Σα ε, βεβαιώ, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι έχετε κάθε ελεύθερο να καταθέσετε όποια ερώτηση θέλετε. Αλλά έχουμε το τρίτο κομμάτι τη ακροασία μα, Μιλή λησμονείτε. Επομένω, όλα αυτά τα ερωτήματα έχουν θέσει στο τρίτο κομμάτι. Να απαντήσει ίσως ο κύριος Λανότ πρώτα για τις ερωτήσεις που τον αφορούν. Καλώς, ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Όσον αφορά τα πιστοποιητικά εκπομπών, δεν είναι πολύ ρευστή η αγορά. Τουλάχιστον όσον αφορά τα χρηματιστήρια που συναλλάσσονται σε αυτά τα πιστοποιητικά. Επομένω, μπορούμε να περιμένουμε ότι θα έχουν την ίδια αντιμετώπιση με τα λοιπά χρηματόγραφα, αξιόγραφα και τις ε, συναλλαγές ενδεχομένω ε, OTC για τον κύριο Γκέμπελς. θα έλεγα προ όλου εκείνου, είτε από το, το χώρο των συναλλαγών, είτε από τι τράπεζε που αμφισβητούν τα στοιχεία για τα OTC, να ρίξουν μια καλύτερη ματιά στα στοιχεία. Γιατί εγώ τα παρακολουθώ εδώ και χρόνια, δεν βλέπω τίποτε λάθο, δεν καταλαβαίνω τι είναι αυτό που αμφισβητούν δηλαδή. Εάν λοιπόν είτε είναι τα χρηματιστήρια, είτε είναι οι επενδυτικέ επιχειρήσει, ε, σε αδυναμία να δώσουν καλύτερα στοιχεία, έστω εντάξει. Γι' αυτό υπάρχει αυτή η νέα μορφή αδειοδότησης έτσι ώστε ο παρέχον της πληροφορίας να επιτρέπει στις αρχές ε, να καταγράψουν επακριβή στοιχεία. Αυτό που έχω ακούσει εγώ σαν δικό στοιχείο είναι το 14 15%. Αυτό μπορώ να προσφέρω στη συζήτηση. Για το OTF, σαν απάντηση στα OTC. Ναι. Για θα μπορούσε όμως να είναι και MTF. Γιατί να δημιουργηθεί μια νέα κατηγορία. Απλώς περιπλέκουμε το έργο του νομοθέτη. Για μένα φαίνεται μάλλον να είναι μεταξύ πολυμερών ε, πλατφορμών συναλλαγών και εσωτερικής συναλλαγής, ε, η συστημικής ε, εσωτερήκευσης, αυτές οι λύσεις. Δηλαδή, πρόκειται για επενδύσεις οι οποίες γίνονται για λογαριασμό κάποιου, αλλά κατά του ίδιου του, του κεφαλαίου. Επομένως δεν βλέπω γιατί δεν μπορεί να θεωρηθεί ω ένα υποκεφάλαιο του MTF. Για τι συναλλαγέ υψηλή συχνότητα, ξέρω επίση ότι είναι μια σύντηση που έχει κρατήσει τουλάχιστον τρία χρόνια και που εν τέλει πιστεύω ότι δεν θα πρέπει και να λησμονούμε πόσα είχε πολύ σημαντικό αντίκτυπο διότι επέτρεψε επενδύσει στη νέα τεχνολογία. Μην ξεχνάμε ότι οι επικρίσει κατά τον Μεφιτή ήταν παλιά, ότι είναι πολύ γραφειοκρατικό και επιβαρύνουν πολύ με γραφειοκρατία όλη τη δικασία. Και όμω επωφελήθηκαν και δει ποιοι η νέα τεχνολογία και δει οι Ηνωμένε Πολιτείε που έχουν πάρα πολύ ε, μεγάλη εξέλιξη στον τομέα αυτό. Επομένω, έχουν μπορέσει να ανταποκριθούν στι προκλήσει, τεχνολογικέ εξελίξει που εμφανίστηκαν στη τελευταία ανάλυση και στι δύο όχθε του Ατλαντικού, αλλά υποφελήθηκαν από τη μια μεριά για αυτόν τον λόγο και μόνο. Εάν χρειαστεί να ρυθμιστεί, εντάξει, αλλά αυτό σημαίνει ότι θέλουμε να ρυθμίσουμε τη λειτουργία της τεχνολογικής εξέλιξης. Αυτό θέλουμε. Δεν ξέρω αν η Επιτροπή λέει ότι ναι υπάρχουν άλλα μέτρα για λειτουργία ή για έλεγχο του, των κινδύνων. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ένα νέο flash crash δεν θα ξαναφανιστεί. Αν θέλετε να αποκλείσετε 100% μια τέτοια, ένα τέτοιο ενδεχόμενο πρέπει απλώς να εμποδίσετε τις επενδύσει στην τεχνολογία. Um, <coughs> uh, για την ερώτηση του κ. Φέρμπερ. Ρευστότητα έναντι αλγορίθμων. Ίσως δεν ήμουν πολύ σαφής σε αυτό που είπα. Συναλλαγές με βάση αλγορίθμους είναι η επικεφαλίδα. Και μετά έχουμε το υποκεφάλαιο που είναι οι συναλλαγές υψηλής τυχνότητας, που πάλι κατανέμονται σε δύο τομείς. Ένα τομέα ο οποίος μπορεί να προσφέρει ρευστότητα, και ένας τρόπος εργασίας των αγορών με, που προσφέρει ρευστότητα και μετά υπάρχει μια άλλη σειρά από τεχνικές που προσφέρουν όγκο αλλά όχι ρευστότητα. Αυτή είναι η διάκριση στην οποία προέβαινα εγώ. Για δε το ενδεχόμενο ενό flash crash, crash απλώς θέλω να εξηγήσω με τον τρόπο αυτό ότι καθώς η μεγάλη πλειονότητα των συναλλαγών υψηλής συχνότητας ήταν μια ευκαιριακή επιλογή. Δηλαδή βλέπω ένα τρένο να περνάει και το παίρνω για να προσπαθήσω να εκμεταλλευτώ μια συγκυρία, να κερδίσω δηλαδή από μια ευρωϊκή συγκυρία. Πρέπει έτσι να αντιμετωπίζονται. Αυτό που κάνει η Επιτροπή όμως είναι ότι ζητώ από τους εναλλασσόμενους σε υψηλή συχνότητα να προσφέρουν ε, ρευστότητα στην αγορά. Δεν έχει καμιά λογική. Μάλλον χρειάζεται μια κάποια προσαρμογή. Όπως και εγώ στο παρελθόν που υπέγραφα συναλλαγές χάραξης αγοράς με συναλλασσόμενους και ήξερα πάρα πολύ καλά ότι αν υπογράφω συμφωνία ρευστότητα, δεν μπορώ και να υποχρεώσω το χρηματοπιστωτικό αυτό οργανισμό 100% ανά πάσα στιγμή και για κάθε περίπτωση να έχει ρευστότητα, γιατί προφανώ δεν μπορούν οι πραγματικέ συνθήκε, ο, ο κόσμο, ε, ο πραγματικό ρεαλιστικό να επιτρέψει μια τέτοια εξέλιξη ένα τέτοιο ενδεχόμενο, αποκλεισμό δηλαδή κάθε κινδύνου. Από την άλλη, εάν θέλουμε αυτός που θα προσφέρει ε, ρευστότητα μάλλον αυτό που συναλλάσσεται σε ψηλή συναλλαγή να προσφέρει εξαπάντως και ρευστότητα, τότε μάλλον οι περισσότεροι θα πούνε «Α, sorry, δεν γίνεται» και οι λοιποί θα το δεχθούν εμένα και θα δεσμευθούν ενδεχομένως νομικά, καθώς είναι και καθήκον τους από ό,τι γνωρίζω τουλάχιστον εγώ, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει μια απόλυτη, ε, έναν απόλυτο αποκλεισμό κάθε κινδύνου. Αυτό πρέπει να είναι ξεκάθαρο. Για δε το προσδιορισμό των τιμών και τη λειτουργία καταγραφή τιμών που ρωτήθηκε από την άλλη πλευρά, όταν λειτουργεί με τόση ταχύτητα το σύστημα, αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλη σημασία. χωρίς να θέλω να προσβάλλω κανέναν, αυτό που ζούμε στην αγορά αυτή τη στιγμή είναι διεστραμμένο. Δηλαδή έχουμε τον γνήσιο επενδυτή, ο οποίος φοβάται ότι κινδυνεύει από, την, ε, από τον επενδυτή υψηλής συχνότητας και χρησιμοποιεί είτε σκοτεινούς χώρους συναλλαγών, σκοτεινό βένιο δηλαδή, είτε OTC προκειμένου να συγκαλυφθεί από αυτόν τον επενδυτή υψηλής συχνότητας για να προστατεύσει την τιμή του προϊόντος. Δηλαδή, κατά κάποιον τρόπο, η σκοτεινή πλευρά της αγοράς εκτρέφει την συναλλαγή υψηλής συχνότητας και τούμπαλη. Γι' αυτό πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Γιατί η σκοτεινή όψη της αγοράς, θα έλεγα, εκτρέφεται εις βάρος της φωτεινής πλευράς της αγοράς τις ανοιχτής δηλαδή συναλλαγές Και όποτε μιλούμε με τους ε, παράγοντες αγοράς, ε, μας μιλάνε για έξυπνο χρήμα και για ανόητο χρήμα. Το ανόητο χρήμα το εντοπίζουν στη φωτεινή πλευρά της αγοράς και το έξυπνο στη σκοτεινή. Αυτό λοιπόν εμένα με προβληματίζει ιδιαίτερο. Δεν μπορεί κανείς δηλαδή να λέει ότι η σκοτεινή πλευρά είναι η ευφυής πλευρά και η φωτισμένη είναι η ανόητη. Θέλετε να πείτε τίποτα για το OTF, το σχόλιο αυτό. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Πολύ καλή ερώτηση για το OTF. Δεν είμαι σίγουρος ότι θα προσφέρουν κάτι τα OTF και συμφωνώ με τον προλαλήσαντα. Μάλλον και επιτρέψτε μου παρεμπιπτόντως, γιατί δεν θέλω να επισέλθω πολύ, αλλά στο θέμα της αγοράς των over-the-counter, τα ποσοστά, τι να σας πω, η Thomson Reuters δίνει το 40% ως ποσοστό, θεωρείται αξιόπιστη πηγή, αλλά και 15 να είναι και 20 να είναι. Μάλλον 14% δίνει και μπορεί να είναι και 15 και 20, αλλά εν πάση περιπτώσει μιλάμε για OTC και για OTF. Πολύ καλά. Ας δούμε λοιπόν το OTF ως εφεύρεση τι προσφέρει επιπλέον στη συζήτηση. Δεν νομίζω ότι μας προσφέρει τίποτα. Ιδιαίτερα πλεονεκτήματα. Αυτό λοιπόν που πρέπει να κάνουμε θα είναι να ενισχύσουμε τον ορισμό του OTC στο MIFID. Ο ορισμός, λέει, ο ορισμός της ε, OTC είναι μάλλον αδύναμος, αν υπάρχει. Είναι το 53 μόνο εδάφιο και αυτό που λέει βασικά είναι ότι αφορά συναλλαγές που ξεπερνούν τα μεγέθη της αγοράς. 48% είναι κάτω από το, τα μεγέθη της αγοράς, το είδαμε και με πολύ αξιόπιστη έρευνα ως πηγή. Και άρα και πάλι αντι, ε, αντιπαρέρχεται, μάλλον το πνεύμα της ΜΥΦΙΝΤΕΝΑ. Άρα αυτό που θέλουμε είναι να ενισχύσουμε τον ορισμό του OTC. Και δεν είμαι πεπισμένος ότι αν αυτό δεν γίνει, αν δεν ενισχυθεί αυτός ο ορισμός, μπορούμε να ρυθμίσουμε το παραμικρό με, έναν καλύτερο ορισμό και τα OTF δεν χρειάζονται στη τελευταία ανάγνωση. Ευχαριστώ κύριο Σμιτ εκ μέρου των Φιλελευθέρων και μετά κυρία Σουίνμπερν εκ μέρου τη ΕΣΥΑ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ πολύ τους προσκεκλημένους μας για τις δύο πρώτες παρεμβάσεις τους. Δεν είναι και πολύ εύκολο να τα καταλάβει κανείς όλα αυτά. Ένας από τους ομιλητές είπε ότι είναι στρεβλωμένη αγορά λίγο πολύ, ο άλλος είπε ότι λειτουργεί καλά. Οπότε, ρωτάω τον κύριο Λανουά. Εσείς πιστεύετε ότι υπάρχει κίνδυνος υπερβολικής ρύθμισης και κατάλαβα καλά, λέτε ότι ίσως το κύριο πρόβλημα με την σημερινή οδηγία MIFID είναι η έλλειψη της καλής της εφαρμογής Δηλαδή ότι θα μπορούσαμε ήδη να τα είχαμε κάνει αυτά που πρέπει να κάνουμε, τα κράτη-μέλη δηλαδή. Σας καταλαβαίνω καλά. Και για σας κύριε Φιλιππονά, εσείς πώς ορίζετε τα κριτήρια για τις υψηλής συχνότητα συναλλαγές. Γιατί νομίζω ότι είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό. Ξέρετε την ιστορία για το Σπιν Γιάννη. Ήτανε, έπρεπε να καταστραφεί, αλλά τελικά δεν λειτουργήσε. Οπότε εμεί πώς χρησιμοποιούμε την τεχνική. Δεν θα έπρεπε να την χρησιμοποιούμε για τους στόχους μας. Και δεν είναι ρητορική η ερώτησή μου. Κοίταξτε, εγώ είμαι φιλελεύθερος και νομίζω ότι η τεχνική είναι κάτι πολύ χρήσιμο και έχει αποδειχτεί η χρησιμότητά της. Ήδη από τον 17ο αιώνα είχαμε πει ότι όλα τα έχουμε βρει. Όχι, δεν τα είχαμε βρει όλα και όσο προχωράμε όλο και περισσότερα πράγματα βρίσκουμε και όλο και περισσότερες τεχνικές που θα μπορούσαμε κάλλιστα να τις χρησιμοποιήσουμε για να βελτιώσουμε την κατάσταση αντί να την μπλοκάρουμε. Αυτή είναι η ερώτησή μου για σας και για τους δύο τώρα. Έρχομαι στη διαφάνεια. Εγώ βεβαίω και θέλω τη διαφάνεια. Από το 1766 την έχουμε εμεί. Αλλά Μήπως τελικά δεν είναι αυτό που χρειάζεται η πάρα πολύ μεγάλη διαφάνεια για την καλή λειτουργία. Μήπως δεν θέλουν όλοι να γνωστοποιούν τα πάντα όταν θέλουν να κάνουν μια συναλλαγή. Το είπατε κι εσείς, άνθρωποι είμαστε όλοι. Και έχω και μια γενική ερώτηση που δεν ξέρω αν εμπίπτει σε αυτό το πλαίσιο. Επί την Deutsche Börse και την Euromex ε, μιλάμε για συγχώνευση και το εξετάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τώρα. Εσείς πιστεύετε ότι κάτι τέτοιο πώς, τι αντίκτυπο θα έχει στην αγορά, θα δημιουργήσει μεγαλύτερο μονοπόλιο στην Ευρώπη. Ίσως βέβαια να εμπίπτει στο τελευταίο τμήμα της ακορασής μας, αλλά εγώ δυστυχώς πρέπει να φύγω, δεν θα μείνω εδώ μέχρι το τέλος. Και νομίζω ότι αυτό το θέμα είναι πολύ σημαντικό, γιατί είναι κάτι που συμβαίνει τώρα. Όταν ξεκινήσαμε με την οδηγία MIFID, κύριε Πρόεδρε, ήταν για να ανοίξουμε την αγορά, για να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια, για να προστατεύουμε τον επενδυτή. Αναφερόταν και η φιλελευθεροποίηση, αλλά εντάξει, τόσο δεν θα το αναφέρω σαν όρο τώρα, γιατί θεωρείται κακιά λέξη. Τώρα μιλάμε για κατακαιρματισμό. Για μένα, ο κατακαιρματισμός μπορεί να σημαίνει επιλογές για τους ιδιώτες και χαμηλές τιμές για υψηλή ποιότητα. Ευχαριστώ. Η κυρία Σούιμπερκ. Ευχαριστώ. Η ουσία απαντήθηκε κάπως, αλλά εγώ θα περάσω από τις σημερινές τάσεις και θα προσπαθήσω να ακούσω όσο γίνεται περισσότερα πράγματα από τους ειδικού. Προσπαθώ να δω κατά πόσο οι δύο πυρογνώμονες που έχουμε εδώ σήμερα πιστεύουν ότι η ευρωπαϊκή αγορά κεφαλαίων και για το χρέος και για τις μετοχές εξυπηρετούν τους στόχους και κατά πόσο οι προτινόμενες αλλαγές στο κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κάνουν αρκετά πράγματα για να ενισχύσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση και την αξία των συναλλαγών, των ευρωπαϊκών δηλαδή συναλλαγών με τα επιπλέον μέτρα. Ενθαρρύνονται οι αγορέ. Αυτό ξέρουμε ότι έχει μεγάλη σημασία για την οικονομική μας ανάπτυξη που δεν πάει και τόσο καλά τώρα. Τότε και για το κόστος των επενδύσεων, ιδιαίτερα όσον αφορά τους επενδυτές μακροπρόθεσμα. Με την εφαρμογή της ΜΥΦΙΤ είδαμε ότι μειώνεται το κόστος των συναλλαγών, αλλά από την άλλη με τα συναλλαγματικά ε, διαπιστώνουμε ότι είναι αλλιώς τα πράγματα. Οπότε τι μέτρα θα έπρεπε να ληφθούν με την οδηγία MIFID ή με άλλα νομοθετήματα έτσι ώστε να έχουμε πραγματικά ένα προ και μετά συναλλακτικό περιβάλλον ευνοϊκό. Ποιος θα ξεκινήσει πρώτα, μήπως ο κύριος Φιλιππονά πρώτα. Ευχαριστώ. Ακόμα ναι. γράφω εδώ τις ερωτήσεις σας. πώς να καθορίσουμε ε, κριτήρια για το over the counter, για τις εξωχρηματιστηριακές ε, συναλλαγές. Για τις ε, συναλλαγές υψηλής συχνότητας. Είναι ένα μέσον, αλλά όταν πάμε στις οικονομικές αγορές δεν είναι ο στόχος. Δηλαδή, ο στόχος της οδηγίας MIFID είναι να εξυπηρετήσει την οικονομία, να προστατεύσει τον καταναλωτή με δύο λόγια και όταν η τεχνολογία μπορεί να βοηθήσει σε αυτό, εντάξει η τεχνολογία φυσικά και είναι κάτι που πρέπει να προωθούμε, να αναπτύσσουμε, είναι κάτι θαυμάσιο. Ο στόχος πάντως είναι πρώτον και κατά κάποιο τρόπο για να απαντήσω και στις άλλες ερωτήσεις, το δεύτερο γύρο ερωτήσεων, ε, Εξυπηρετούμε το στόχο αύξησης κεφαλαίου, εξυπηρετούμε τους επενδυτές που θέλουν διαφάνεια και ε, δικαιοσύνη, έτσι ώστε να είναι σίγουροι ότι τα κεφαλαία τους εξυπηρετούν την πραγματική οικονομία. Κατά πόσο βοηθάει, βοηθούν οι ε, υψηλές συχνότητες συναλλαγές. Νομίζω ότι οι πολιτικοί πρέπει να αναρωτιούνται. Βοηθάει ή δεν βοηθάει. Μερικές φορές όμως η απάντηση είναι ναι και άλλες φορές η απάντηση είναι όχι. Όταν ερχόμαστε τώρα στο OTF, είναι δύσκολο εδώ να υπολογίσουμε το νόγκο, όπως επίσης και για τις ε, υψηλές συχνότητες σε συναλλαγές. Είναι δύσκολο. Εξαρτάται από τις τάσεις. Άλλοτε υπάρχει μια τάση και διαπιστώνουμε ότι υπάρχει μεγάλος όγκος, άλλοτε όχι. Και από αυτό δεν εξυπηρετείται η οικονομία. Το ότι χρησιμοποιείται ε, ιδιαίτερα προηγμένη τεχνολογία για μένα είναι κάτι ουδέτερο. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι καλό ούτε ότι είναι κακό. Το θέμα είναι το χρειαζόμαστε ή όχι. Αυτή είναι η δικιά μου πεποίθηση. Παρέμβαση εκτός μικροφώνου από τον κύριο Σμιτ. Αν το χρειαζόμαστε, την τεχνολογία χρειαζόμαστε όσο γίνεται πιο προηγμένη τεχνολογία όταν αυτή εξυπηρετεί την οικονομία. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου υπάρχει υπερβολικά μεγάλη διαφάνεια. Άμα θέλετε να συναλλαχθείτε για το 2% των τίτλων μιας ε, εταιρείας, εντάξει δεν μας ενδιαφέρει. Αλλά το θέμα είναι ότι οι περισσότερες εξοχρηματιστηριακές ε, συναλλαγές είναι μεγάλο όγκου. Ε, μίλησα με ένα χρηματιστή, ο οποίος μπορεί να μην γνωρίζει πολύ καλά την οδηγία, αλλά τι μου λέγε. Μου λέγε, ότι οι 300 500 ευρώ είναι οι μεγάλες ποσότητες βάσει της οδηγίας Μίδιτ. Είναι αυτές μεγάλες ποσότητες, μεγάλα ποσά. Πολλά εκατομμύρια ευρώ είναι κανονικά σε τίτλους. Οπότε βέβαια και υπάρχει όριο στην ε, διαφάνεια. Μερικές φορές πρέπει να είμαστε διακριτικοί. Αλλά όταν έχουμε μεγάλο όγκο που όμως περνάει από τους μηχανισμούς ε, μικρών ε, ε, ποσών, τότε τα πράγματα στρεβλώνονται γιατί στον πραγματικό κόσμο δεν ισχύει ο ίδιος ορισμός. Ρωτήσατε κάτι και για τα μονοπόλια. Α, για τη συγχώνευση, ναι. Θα μπορούσα να μιλήσω γι' αυτό αν θέλετε, αλλά πιστεύω ότι είναι κάτι διαφορετικό και πιστεύω ότι δεν είναι ένα θέμα που έχει να κάνει με αυτό που συζητάμε σήμερα. Δεν νομίζω ότι είναι δικιά μας αποστολή να σχολιάσουμε για αυτή την περίπτωση. Δεν είμαι πεπισμένος. Ο κύριος Λανουά. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω και εγώ και να είμαι σύντομο. Πρώτα απ' όλα για την υπερβολική ρύθμιση. Ε, εξαρτάται πώ μετράει κανεί την υπερβολική ρύθμιση. Αν δούμε την οδική και συγκρίνουμε με την MIFID 1, νομίζω ότι είναι παραπάνω 50%. Αν δούμε τον αριθμό των άρθρων, των ε, εκτελεστικών μέτρων, ε, πρόκειται για 20 εφαρμοστικά μέτρα, τώρα έχουμε τις ε, πράξεις που είναι 50. Άρα υπάρχει νέα ρύθμιση. Αν όμως δείτε στο σύνολό του το κείμενο, δεν διαφέρει τόσο πολύ από το μη φιντενα. Προσθέτει κάποια πράγματα, κάνει κάποιες διευκρινήσεις, οπότε δεν θα έλεγα ότι πρόκειται για υπερβαλλική ρύθμιση. Διευκρινίζει το τι ήτανε, ε, φτιάχνει νέες κατηγορίες για τα ΟΤΕΦ και μιλάει και για τις ε, μετασυναλλακτικές ε, πληροφορίες. Πριν μιλούσε μόνο για πριν το διακανονισμό. Συμψηφισμός στα, στις δύο φάσεις. Είναι δύσκολο λοιπόν να το απαντήσουμε αυτό ακριβώς, αλλά πιστεύω ότι έχετε δίκιο γιατί ότι μετά από τέσσερα χρόνια να κάνουμε μια αναθεώρηση ήδη είναι δύσκολο. Θα ήμουν πολύ προσεκτικός. Τώρα κάτι και για την Κομισιόν που έχει κάποια πολιτική χρειά. Μερικές φορές δεν καταλαβαίνουμε και οι κυβερνήσεις ε, μερικές φορές για μερικά πράγματα λένε ότι είναι θέμα κοινή λογικής, αλλά μερικές φορές μπαίνουν κάποια πράγματα απλώς και μόνο για να κοπνοποιηθούν κάποιες ομάδες. Ότι κοιτάξτε, εμεί ασχολούμαστε με αυτό που θέλετε. Τώρα για τη διαφάνεια, κατά πόσο έχουμε υπερβολική διαφάνεια. Είναι πολύ δύσκολο να πούμε πως υπάρχει υπερβολική διαφάνεια. Κυρίως να το πεις αυτό σε κάποιον που δεν είναι μοιημένος. Ακούγεται πολύ περίεργα. Προφανώς ο κόσμος θέλει 100% διαφάνεια, αλλά εμείς ξέρουμε ότι με τη νέα ε, πρόταση, ορισμένοι δεν θέλουν 100% διαφάνεια. Υπάρχει κάποια αλλαγή πλεύσης και εξηγείται στις αγορές και γι' αυτό έχουμε και τις εξοχρηματιστηριακές συναλλαγές, γιατί ορισμένοι θέλουν οι συναλλαγές εκεί να γίνονται διαφορετικά. Τώρα η Deutsche Börse και το χρηματιστήριο του New York, το Next, η συγχώνευσή τους. Αυτή η ερώτηση εγώ πιστεύω ότι έχει να κάνει με το θέμα μας. Έτσι δημιουργείται περισσότερο μονοπόλιδες πώς θα θέσει. Πιστεύω ότι έτσι θα έχουν πολύ σημαντικό ρόλο να παίξουν ε, στον ε, διακανονισμό και συμψηφισμό. Αλλά εξαρτάται ποια αγορά κοιτάς. Κοιτάς την αγορά της Ευρώπης ή του κόσμου. Εμείς βέβαια, από τη δικιά μας την πλευρά, θα πούμε όχι. Τώρα, τέλος, για την ερώτηση του κατά πόσο κάνουμε αρκετά πράγματα με την πρόταση αυτή προκειμένου να υπάρχει χρηματοδότηση στην πραγματική οικονομία. Για μένα το μεγαλύτερο πρόβλημα εδώ και που δεν βρίσκει λύση στην οδηγία αυτή είναι πώς επιτρέπουμε σε ορισμένους μικρούς να έχουν πρόσβαση στην χρηματοδότηση. Γιατί μερικές φορές η μόνη χρηματοδότηση που έχουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι οι τράπεζες. Ενώ ίσως θα έπρεπε να μπορούν να έχουν και πρόσβαση στις κεφαλαιογορές. Η πρόσβαση έχει μειωθεί στις σκανδιναβικές χώρες, στις χώρες Benelux επιτρέπουν ένα είδος πρόσβαση. Και με την κρίση έχει μειωθεί η πρόσβαση στη χρηματοδότηση. Τι κάνουμε με την οδηγία αυτή. Μπορούμε να ξαναδούμε το άρθρο αυτό για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά υπάρχουν και άλλα πράγματα όπως είναι η οδηγία για τη διαφάνεια, που δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Τι άλλα μέτρα θα έπρεπε να λάβουμε υπόψη μας για να ενισχύσουμε αυτή τη τάση, να ενισχύσουμε τον ανταγωνισμό στις τράπεζες, δηλαδή να επιτρέψουμε περισσότερο επίσης όρις πρόσβαση στις ε, ε επιχειρήσεις ώστε να έχουν πρόσβαση εξίσου στο κεφάλαιο. Θα έπρεπε λογιστικέ προδιαγραφέ να μειωθούν, τα κριτήρια δηλαδή για τι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Είναι δύσκολο να απαντήσει κανεί αυτό. Ωραία, έχω ακόμα δύο ερωτήσεις σε αυτό το γύρο, μία από τον κύριο Κάφα και μία από τον κύριο Τούτα. Ε, κύριε Κάφα. Ναι. Μία ερώτηση γενικής φύσεως προ τους ομιλητές ε, σε σχέση με τη σωστή ισορροπία, σύμφωνα με την απόψή τους, ε, μεταξύ του ανταγωνισμού και μιας μορφής συγκέντρωσης που νομιμοποιείται από το γεγονός ότι οι αγορές εξορισμού ακόμη και από το μεσαίωνα αγορά είναι ο τόπος όπου συναντιέται η προσφορά με τη ζήτηση. Αν έχουμε πολλές αγορές τέτοιου τύπου όπως συμβαίνει σήμερα έχουμε κατακαιρματισμό, έχουμε πολλαπλές τιμές και συνεπώς αύξηση του κόστους για τους χειριστές, για τους διαχειριστές. δεν μιλάμε φυσικά εδώ για ένα πανευρωπαϊκό ενιαίο χρηματιστήριο. Πώς θα Μιλάμε για το πώς θα βρούμε την ισορροπία μεταξύ των διαφόρων περιπτώσεων ώστε να έχουμε την απαραίτητη τη εξυπηρέτηση αλλά και την ε, ικανοποίηση του στόχου ε, ουσιαστικά συνύπαρξης όλων των διαχειριστών. Δεν ακούγεται μετάφραση στα αγγλικά. Αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, κάποιο ήχος από την καμπίνα. Τα γερμανικά λειτουργούν. Ναι. Θέλετε να μιλήσετε γερμανικά την επόμενη φορά, πάντα ο μιλητής. Λοιπόν, η πρώτη ερώτηση, δεν ξέρω αν την άκουσαν οι ομιλητές. Ε, Ποιο είναι ο σωστός βαθμός ισορροπίας μεταξύ αυτών των δύο λειτουργιών. Το δεύτερο στοιχείο αφορά τις συναλλαγέ υψηλή συχνότητα. Έγιναν πολλές επενδύσεις, Μα το υπενθύμησαν αυτόν, ωστόσο αυτές οι επενδύσεις ήταν αποδοτικές. Πιστεύω ότι ως νομοθέτες θα πρέπει να πούμε ότι αν χρειαστεί να επανέλθουμε σε άλλους ε, κανόνες λειτουργίας, ε, έχουμε δημιουργήσει κανόνες, έγιναν επενδύσεις, έφεραν τις αποδόσεις τους, ε, τα κέρδη που προέκυψαν. Μπορούμε λοιπόν να αλλάξουμε τους κανόνες, αυτό μπορούμε να το κάνουμε νόμιμα το επιχείρημα ότι έχουν γίνει επενδύσεις ε, με κάποιο κόστος και δεν μπορούμε να αλλάξουμε τους κανόνες δεν είναι αποδεκτό σήμερα. Όσον αφορά τώρα τι συναλλαγέ, ε, υψηλή συχνότητα, έχει πραγματοποιήσει η Finance Watch μελέτη, ή προβλέπει τέτοιε μελέτε για να γνωρίζει ποιο κέρδισε και ποιο έχασε σύμφωνα με τις συζητήσεις που έκαναμε ορισμένα σε επενδυτικές εταιρείες έχουν την εντύπωση ότι επειδή είναι πιο αργή από του, όσους πραγματοποιούν συναλλαγές υψηλής κοινότητας θεωρούν ότι είναι μόνιμα αποκλεισμένοι από την αγορά. Υπάρχει λοιπόν η δυνατότητα εξισορρόψης των κερδών ορισμένων και των απολειών ορισμένων άλλων. Και η τελευταία ερώτηση σχετίζεται, δεν ξέρω αν ο κ. Φιλιππονάρτο έχει ήδη απαντήσει ή όχι, αν το έχει απαντήσει με συγχωρείτε που επαναλαμβάνω. Η τρίτη μου ερώτηση λοιπόν είναι η σαφής διάκριση μεταξύ της, ε, των ε, καλών συναλλαγών και των ε, υψηλής συχνότητας και των κακών. όπου τα κακά εντός αγωγικών χρήματα διώκουν τα καλά εκδιώκουν ουσιαστικά και προκαλούν ολίσθηση των ε, ε, κεφαλαίων αγορών προς ε, μια μορφή καζίνο αντί να πληρούν την, τον αρχικό τους ρόλο. Κύριος Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ο εισηγητή μας είπε ξεκινώντα ότι υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για μια γενικότερη ρύθμιση. Ο κύριος Σμιτ μας είπε ότι στη συζήτηση προκύπτει πολύ γρήγορα το συμπέρασμα ότι μπορεί να έχουμε, μπορεί να έχουμε υπερβολική ρύθμιση. Εγώ από, τις, ε, από την εμπειρία που έχουμε και στη δική μου την πατρίδα βλέπω ότι ίσως δεν είναι σωστό τα πάντα να υπαχθούν στα μεφίτς. Δεν είναι αυτό η λύση δηλαδή. Ε, δεν είναι λύση το μύφιτ για να εξασφαλίσουμε έλεγχο και διαφάνεια παντού αλλά για τα πιστοποιητικά των εκπομπών που λέτε ότι δεν επηρεάζουν, ε, δεν θα έπρεπε να υπάρχουν στα μύφιτς. Και ρωτώ τους δύο ειδικούς μας πώς κρίνουν την κατάσταση. Θεωρούν ότι είναι χρήσιμο να επιτρέπονται ενίοτε παρεκκλήσεις ή απλώς θα λέμε όχι αποκλείεται, δεν έχει νόημα να υπάρχουν ε, παρεκκλήσεις. Και για τους δύο απευθύνεται η ερώτηση, λέει η Μακάρτη, ναι. Πρόεδρε. Να ξεκινήσουμε από εσάς. Ε, εκτός μικροφώνου η Πρόεδρος. Η συζήτηση αφορά τον ανταγωνισμό, τα μονοπόλια και τη φυσική ισορροπία για τις αγορές. Είναι δύσκολο να πούμε κάτι. Ίσως συμφωνώ με το διπλανό μου ότι τα κόστη συναλλαγών μειώθηκαν. Δεν γνωρίζω το συνολικό μέγεθος του κόστους. Εφόσον υπήρξε μείωση, πέτυχε ο ανταγωνισμός. Δεν είχε γίνει κάποια συμφωνία, αλλά σύμφωνα με τα δικά μας δεδομένα μας δείχνουν ότι υπήρξε μείωση. Συνεπώς ήταν εποφελές το ότι είχαμε μεγαλύτερο ανταγωνισμό παρότι πολλές εταιρείε το 2005-2006 είπαν ότι όλες αυτές οι επενδύσει είναι υπερβολικά πολλές και η FSA έκανε μια εκτίμηση του κόστου τη μεθόδου υλοποίηση. Ε, μίλησε για πολλά δισεκατομμύρια, αλλά ακόμη και τότε καταφέραμε να παραμενούμε ανταγωνιστικοί, να βελτιώσουμε την ανταγωνιστικότητά μας. Ουσιαστικά το ζήτημα είναι τι βαθμό ανταγωνισμού θέλουμε αλλά ξεκινώντας από το 2001 όταν ξεκινήσαμε την ISD υπήρχαν πάρα πολλά μονοπόλια ενώ σήμερα έχουμε πολύ περισσότερο ανταγωνισμό όχι πλήρη ανταγωνισμό επειδή τα περισσότερε blue chips ε, ε, η συναλλαγή τους γίνεται στις ε, οικίες αγορές τους μπορούμε να κάνουμε κάποια πράγματα και από αυτή την άποψη όσον αφορά τις συναλλαγές υψηλού συχνότητας κατά πόσο πρέπει να υπάρχουν κανόνες λειτουργίας και πάλι ήθελα να πω απαντώντας την ερώτηση του κυρίου Γκέμπελς ο καθορισμός τιμής παρεμποδίστηκε όπως φαίνεται όχι όλες οι ακαδημαϊκές μελέτες μέχρι σήμερα δείχνουν ότι ακόμη και με τις τεράστιες επενδύσεις ο καθορισμός τιμής βελτιώθηκε Ωστόσο, χρειάζεται να έχουμε λειτουργικού κανόνες σε αυτές τις εταιρείε που ασχολούνται με τι συναλλαγέ υψηλού κινδύνου, ώστε να μην υπάρχουν ε, ε, διαταραχές προς την αγορά. Αυτό προτείνεται στη δεύτερη εκδόση της MIFID. Ποιος κέρδισε και ποιος έχασε από όλα αυτά. λαμβάνοντας υπόψη τη μείωση του κόστου συναλλαγών ακόμη και με τους μικρότερους όγκους ε, ως αποτέλεσμα της κρίσης πρέπει να ρίξουμε ματιά στα στατιστικά στοιχεία ε, των ε, χρηματαγορών να δούμε ότι και οι όγκοι και τα κόστη μειώθηκαν η μείωση αυτή του κόστου σημαίνει ότι υπήρξε υγιής ανταγωνισμός ποια είναι η καλή και κακή μορφή των συναλλαγών υψηλής συχνότητας δεν το γνωρίζω. Για την τελευταία ερώτηση, κατά πόσα όλα πρέπει να καλύπτονται από την MIFID, έχω την εντύπωση ότι η MIFID προσπαθεί να επεκτείνει το πεδίο εφαρμογή τη, την αδειοδότηση των trade offenders, ξέρετε ότι είναι κάτι καινούριο. Έχουν γίνει τρεις προτάσεις από την Επιτροπή. Επίσης, όσον αφορά τις συναλλαγές για εκπομπές, ε, δεν έχω κάποια άποψη. Γι' αυτό, όταν επανεξετάζεις κάτι, ε, θέλεις φυσικά να προσθέσεις στοιχεία, ώστε να εξηγήσεις για ποιο λόγο το επανεξετάζεις. Ευχαριστώ. Θα απαντήσω στα γαλλικά, εάν δεν σας ενοχλεί. Εξισορροπία μεταξύ συγκέντρωσης και ανταγωνισμού είναι σαφές ότι ο ανταγωνισμός έχει πολλά πλεονεκτήματα. Επιτρέπει να, γίνει, να υπάρξει πίεση για να είμαστε πιο αποδοτικοί και λιγότερο ακριβοί. Είναι αλήθεια ότι τα κόστη συναλλαγών έχουν χαμηλώσει, ωστόσο αυτό δεν έφτασε μέχρι τους τελικούς επενδυτές ή τουλάχιστον όχι εξ ολοκλήρου. Σε κάθε περίπτωση το κόστος έχει μειωθεί, οι τιμές αυτό αποτελεί ένα άλλο θέμα. Υπάρχουν τα υπέρ και τα κατά, δημιουργήσαμε ένα κατακαιρματισμό που πολλές ε, μελέτες έδειξαν ότι παρά τη μείωση των τιμών χάρη σε διάφορα τεχνολογικά μέσα τις επανευθυγραμμίζουμε. Πιο ουσιαστικό θέμα είναι ότι όταν ξεκινάμε από την αρχή ότι ο ανταγωνισμός έχει πλεονεκτήματα και αυτό είναι αναμφισβήτητο το θέμα είναι να ρυθμίζεται ο ανταγωνισμός αυτός επαρκώς. Αυτό μου κάνει εντύπωση σήμερα είναι ότι σε διάφορες αγορές δεν υπάρχουν ίδιοι περιορισμοί όσον αφορά τη ρύθμιση. Καλό λοιπόν ναι, να υπάρχει ο ανταγωνισμός, αλλά πρέπει να γίνεται με ίσους κανόνες. Πιστεύω ότι αυτό είναι θεμελιώδης σημασία. Διότι όσον αφορά την επιτήρηση αγορών, υπάρχουν αγορές που ε, ρυθμίζονται πολύ περισσότερο από ό,τι άλλες. Η επιτήρηση λοιπόν των αγορών είναι αυτό που ε, σχετίζεται άμεσα με την κατάχρηση των αγορών. Εάν δεν επιβάλλουμε τους ίδιους κανόνες σε όλους, θα υπάρχει διαστρέβλωση του ανταγωνισμού. Συμφωνώ λοιπόν να υπάρχει ανταγωνισμός, αλλά με ίσους κανόνες. Ε, ε, αυτό το επιχειρήματα μπορούμε να τα εξετάσουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό. Με ρωτήσαν τι κάνουμε με την πραγματική οικονομία, κατά πόσο μπορεί να χρηματοδοτηθεί από εδώ. Θα πρέπει όλες οι αγορές Ξέρουμε ότι τα παραδοσιακά χρηματιστήρια επιτελούν ε, τη λειτουργία IPO, Initial Public Offering, το να επιτρέψουν την εισαγωγή νέων επιχειρήσεων στο χρηματιστήριο. Δεν μπορούμε να επικεντρωθούμε μόνο στο ε, δευτερογενή συναλλαγή των blue chips. Ναι, λοιπόν, στον ανταγωνισμό, αλλά ισορροπημένο ανταγωνισμό με ίσους κανόνες. Κατά πόσο η Finance Watch έχει εξαγάγει μελέτη για τους ποιος, και, ποιος κέρδισε και ποιος έχασε, όχι. Αν θα την κάνουμε στο μέλλον θα ήταν μια πολύ καλή ιδέα από τεχνική άποψη. Δεν είναι κάτι απλό να βρούμε τις στατιστικές πληροφορίες για κάτι τέτοιο. Καλό θέμα είναι. Καλό θα ήταν να κάνουμε μια σοβαρή μελέτη επί του θέματος. Μόνο αυτό μπορώ να σας πω αυτή τη στιγμή. Διάκριση μεταξύ των καλών εντό εισαγωγικών και κακών συναλλαγών υψηλού συχνότητα. Ε, ποιο είναι το κομμάτι των συναλλαγών. Ουσιαστικά υπάρχουν δύο τύποι ρευστότητα σε μία χρηματαγορά. Είτε ένα τελικό επενδυτή, συγγνώμη, ένα πραγματικό επενδυτή που θέλει να πουλήσει, συναντά έναν πραγματικό επενδυτή που θέλει να αγοράσει, αυτό αποτελεί ρευστότητα όταν αυτοί οι δύο συναντώνται. Η δεύτερη περίπτωση είναι οι market maker οι οποίοι κάνουν προσφορές ε, με τιμές αγοραστών και ε, πολιτών ε, σε μια αγορά. Πρόκειται για ένα χρήσιμο σύστημα που φέρνει ρευστότητα και που έχει υπόκειται σε κάποιους περιορισμούς. Αυτοί οι δύο τρόποι υπάρχουν για τη δημιουργία ρευστότητας. Οι συναλλαγές υψηλής συχνότητας είναι πραγματικοί επενδυτές, όχι. Ένας άλλος τρόπος δημιουργίας ρευστότητας είναι να έχουμε market maker και εδώ απαντάμε και στο ερώτημα για την τεχνολογία. Μάλιστα η τεχνολογία θα επιτρέψει να κάνουμε market making μόνιμα, δηλαδή προσφέροντας μία τιμή αγοραστή και μία τιμή πολιτή σε ένα χρηματοοικονομικό μέσο για να δημιουργήσουμε ρευστότητα, τότε αυτή η τεχνολογία είναι καλή, διότι διεξάγει μία σωστή συναλλαγή υψηλή συχνότητα. Πρόκειται για προηγμένη τεχνολογία, η οποία έχει νόημα γιατί συμβάλλει στην οικονομία. Όσον αφορά το την ερώτηση του κατά πόσο πρέπει να υπάρχουν εξαιρέσει ε, για τι ε, συναλλαγέ, ε, για τι εκπομπέ. Μια πολύ ειλικρινή απάντηση είναι ότι δεν έχω ψάξει ιδιαίτερα το ερώτημα. Διαισθητικά είμαι λίγο διστακτικός προς κάθε αίτηση εξαίρεσης Ωστόσο, επειδή δεν έχω εμφαθύνει στο θέμα, θα είμαι προσεκτικό στην απάντησή μου. Δεν μου αρέσει να δίνω απαντήσεις που δεν βασίζονται σε κάποια μελέτη. Σα προτείνω να το μελετήσουμε λοιπόν το ζήτημα και να επανέλθουμε σε αυτό το ερώτημα μόλις θα έχουμε το χρόνο. Ευχαριστώ. Περνάμε στο δεύτερο τώρα που αναφέρεται στην προστασία του επενδυτή. από το μη Φιντένα την πρώτη οδηγία και μετά. Ε, πρώτο μιλήτρια είναι η κυρία Βερένα Ρος, που είναι εκτελεστική διευθύντρια της ε, Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ τον εισηγητή καθώ και του βουλευτέ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ευκαιρία που μου δίνει να μιλήσω για το τόσο σημαντικό αυτό θέμα σήμερα. Η αναθεωρημένη MIFID προσπαθεί να ενισχύσει την προστασία των ε, επενδυτών ε, με σαφέστερη, σαφέστερο προσδορισμό των όρων ε, παροχής των υπηρεσιών αυτών. Οι προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής επιτρέπουν να προχωρήσουμε προς ένα αρμονισμένο πλαίσιο πολύ πιο οργανωμένο από αυτό το οποίο έχει προτείνει η MIFID και γνωρίζουμε ότι η MIFID 2 μπορεί να προσφέρει περισσότερα ακόμα ωφέλη. Μια και δεν έχουμε πολύ χρόνο σήμερα, θα ήθελα να επικεντρωθώ σε πέντε τομείς όπου θεωρώ ότι ε, μπορούμε να προχωρήσουμε περαιτέρω με το μέφετ 2 ε, στην προστασία των καταναλωτών, έστω και αν η αγορά είναι κατακαιρματισμένη. Καταρχάς, ε, οι ΕΑΚΑ και οι Εθνικές Αρχές θα πρέπει να είναι συντονισμένες έτσι ώστε να να παρεμβαίνουν για να προστατέψουν τον επενδυτή σε αγορές ή προϊόντα. Ε, και αυτό νομίζω το κομμάτι που αφορά τα προϊόντα είναι ένα σημαντικό βήμα προόδου και αυτό το καθιστά υποχρεωτικό η κατάσταση που αντιμετωπίζουμε τη σύγχρονη εποχή, τεχνολογικές εξελίξεις, περίπλοκη διαστρωμάτωση των χρηματοπιστωτικών αγορών και το ενδιαφέρον του μικρού επενδυτή για συμμετοχή σε αυτέ τι χρηματοπιστωτικέ αγορέ, γεγονότα τα οποία μα υποχρεώνουν να προσφέρουμε καλύτερη προστασία του επενδυτή. Μια προσέγγιση ισορροπημένη είναι απαραίτητη ασφαλώ, εθνική δηλαδή και συντονισμένη ευρωπαϊκή ανταπόκριση, πράγμα το οποίο μπορεί να σημαίνει ε, σημαντικές προκλήσεις προς την υλοποίηση αυτής της προσέγγισης. Κύρια πρόκληση για την ΕΑΚΑ ασφαλώς είναι ε, ο συντονισμό ενδεχομένων δράσεων που αλαμβάνουν οι εθνικέ ε, εποπτικέ αρχέ, συνεπάγεται ότι θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη η ΑΚΑ συγκεκριμένες ανάγκες που ενδεχομένω λαμβάνουν υπόψη ε, οι οποίε υποκλίνονται οι εθνικέ αρχέ, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει και κάποια άλλα στοιχεία να τα εξετάσει στην ευρωπαϊκή του διάσταση ή πάντως στην υπερεθνική του διάσταση. Δηλαδή η ΑΚΑ θα πρέπει να μπορέσει να συγκεράσει διαφορέ και να εξασφαλίσει συντονισμό ανάλογα με τι ανάγκε, χωρί βέβαια αυτό να αποκλείει και εθνική δράση, πράγμα το οποίο βεβαίω μπορεί εν τέλει να προξενήσει ε, κατακαιρματισμό στις αγορές. Φυσικά αυτό συνεπάγεται ταυτόχρονα και προσδορισμό των εξουσιών και ενώ θέλουμε να έχουμε αρκετέ ε, διασφαλιστικές δικλίδες πρέπει να εξασφαλίσουμε και για την ΕΑΚΑ τη δυνατότητα ταχεία αντίδρασης εφόσον αυτό αποβαίνει προ συμφέρον των επενδυτών. Δεύτερος τομέας, στις προδιαγραφέ καταλληλότητας όπου θεωρούμε πως ε, το ΜΥΦΙ τώρα μπορεί να το στηρίξουν και τον ενισχύσουν δύο επιπλέον τομείς, δηλαδή περισσότερη διαφάνεια ως προς το χαρακτήρα των συμβουλών, αν ανεξάρτητας ή όχι, και δεύτερον, αντιμετώπιση της μεροληψίας της σχετικής, που προκύπτει δηλαδή από την προμήθεια που καταβάλει ο εμπλεκόμενος φορέας. Και αυτό Σημαίνει στην πρώτη περίπτωση ότι στις ανεξάρτητες συμβουλές δεν μπορούν οι ε, διαχειριστές χαρτοφυλακίου και εμπλεκόμενες εταιρείε να λαμβάνουν κάποιο τίμημα από εμπλεκόμενα μέρη. Αυτό σημαίνει ταυτόχρονα ότι Μπορεί αντίστοιχα κίνητρα προ τι επενδυτικέ επιχειρήσει να οδηγήσουν σε στρέβλωση αγορά, ενώ θα μπορούσαν οι σύμβουλοι να εξακολουθούν να λαμβάνουν κίνητρα. Πρέπει να είμαστε σαφεί ώστε να μην οδηγηθεί σε παρερμηνία τη κατάσταση ο επενδυτή. Δηλαδή, θα πρέπει ο επενδυτή να έχει σαφή εικόνα και πιστεύουμε ότι οι προτάσει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθούν να εξεύρουν μια καλή ισορροπία στι ε, διαφορετικέ και αντικρουόμενε ανάγκε στον περίπλοκο αυτό τομέα. Επιπλέον, θα ήθελα να αναφερθώ στο τρίτο θέμα, το οποίο έχει να κάνει με την ενίσχυση του πλαισίου βέλτιστης ε, υλοποίησης, βέλτιστης εκτέλεσης, που δηλαδή βελτιώνει τις συνθήκες ενημέρωσης ε, προς τον πελάτη από τον ε, Σύμβουλο Επενδύσεων και ως προς τον τόπο και ως προς τα δεδομένα που αφορούν τον κάθε τόπο εκτέλεσης για την ποιότητα της εκτέλεσης που είναι πάρα πολύ σημαντικά. Η βελτίωση της ποιότητας των πληροφοριών της ενημέρωσης αυτής δηλαδή είναι ουσιώδους σημασία και πιστεύουμε ότι μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερη διαφάνεια για όλους τους επενδυτές στους τομείς αυτούς και εν τέλει να επιτρέψει στον επενδυτή και τον πελάτη να αντιληφθούν πώς εν τέλει θα εκτελεστούν οι εντολές. Στον τέταρτο τομέα που σημειώνεται βελτίωση είναι ο τομέας που επιτρέπει τη δυνατότητα επενδυτών και επιχειρήσεων από τρίτες χώρες να αναλαμβάνουν τις δραστηριότητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να υπάρχουν σε έναν ενοποιημένο χώρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση κανόνες πρόσβασης, αλλά οι περιορισμοί στην πρόσβαση δεν θα πρέπει να αποκλείσουν κάθε δυνατότητα παρέμβασης ε, χειριστών ε, ε, διαχειριστών καλύτερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ανάληψης δραστηριοτήτων επενδυτικών, γιατί αυτό μπορεί να αποβεί εις βάρος και των επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βέβαια τον αποκλεισμό της αγοράς των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Πέμπτον, καλωσορίζουμε τις, τα συμπεράσματα, τα σχετικά με τα διαστρωματωμένα προϊόντα MIFID, ε, που μπορούν να αποτελέσουν μια καλή λύση σε σχέση με τα παράγωγα επί εμπορευμάτων. Συνεργαζόμαστε στενά με, τους, ε, με τις άλλες ρυθμιστικές αρχές για να βελτιώσουμε την προστασία των καταναλωτών έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε εν τέλει ένα ισότιμο πεδίο ανταγωνισμού μεταξύ των διαφόρων επενδυτικών προϊόντων. Και εν τέλει πιστεύω ότι θα πρέπει να επενθυμίσω πως η MIFID 1 έχει ήδη προσφέρει αρκετούς κανόνες για την προστασία του καταναλωτού. Έχουμε εξασφαλίσει τους τα τελευταία χρόνια κάποια πρόοδο για την προστασία των καταναλωτών, των επενδυτών. Ε, ωστόσο, δεν θα πρέπει μόνο να ασχολούμαστε με τη μεταρρύθμιση των κανόνων, αλλά να επιδιώκουμε την ουσιαστική εποπτεία και εφαρμογή των ισχυών των κανόνων, εφαρμογή και ε, εποπτεία που θα πρέπει να ισχύει εξίσου σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εδώ θα πρέπει να στρέψουμε την προσοχή μα. Σωστή υλοποίηση λοιπόν και εποπτεία υπό την MIFID 1, που στο τελευταίο ένα θα εξακολουθήσει να ισχύει για αρκετό διάστημα, ακόμη και κατά την περίοδο που συνεχίσει η διαπραγμάτευση για την MIFID 2. Η ΑΕΚΑ και η ΣΕΖΑΡ νωρίτερα είχαν κάνει σημαντική, είχαν προσφέρει σημαντική συμβολή ως προς την εφαρμογή των ε, κειμένων της ΜΥΦΙΝΤΕΝΑ. Εμείς πιστεύουμε ότι μπορούμε και από πλευράς μας να συμβάλλουμε αντίστοιχα και για τη ΜΥΦΙΝΤΕΝΑ και για τη ΜΥΦΙΝΤ2 και με την υποστήριξη του Συμβουλίου του Κοινοβουλίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αυτή τη διαδικασία την νομοθετική φυσικά πιστεύουμε ότι θα μπορέσουμε και εμείς να βελτιώσουμε από πλευράς μας κάποιες προδιαγραφές ε, εφόσον βέβαια κρίνει απαραίτητη και παρείται αυτήν την εξέλιξη η νομοθετική αρχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριο Ζουέ από την αντίστοιχη αρχή τη Γαλλία, σα ευχαριστώ θερμά για την διεξοδική απάντηση που δώσατε γραπτό. Τώρα σα καλώ να μιλήσετε μόνο για πέντε λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, κύριε Σιγητά Φερβέρ, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά έχω κάτι γραπτό, το οποίο είναι στη διάθεση των Ευρωβουλευτών. Ε, αυτό που θέλω όμως, μετά τόσα έχουμε ήδη τόσο καλά ακούσει, να υπογραμμίσω ότι το θέμα της αναθεώρησης της οδηγίας είναι κάτι το απλό. Πρώτα απ' όλα θέλουμε να έχουμε αγορές όπου οι τιμές διαμορφώνονται με διαφάνεια προς εξυπηρέτηση της οικονομίας και δεύτερον, δεύτερος στόχος είναι η προστασία όλων των επενδυτών. Για μας ο απολογισμό από την πρώτη οδηγία δεν είναι κάτι τόσο καλό γιατί υπήρξε κατακερματισμός, αδιαφάνεια, έλλειψη ανταγωνισμού ανάμεσα στις αγορές και τις πλατφόρμες. Δεν ελέγχεται καλά το θέμα των συναλλαγών ε, που γίνονται με υψηλή συχνότητα ούτε και το θέμα της προσφοράς ρευστότητας. Όπως υπογραμμίστηκε, ο κατακαιρματισμός οδηγεί σε αδιαφάνεια. Η τεχνολογία και η αδιαφάνεια είναι δύο πράγματα τα το ένα τροφοδοτεί το άλλο. Οι επενδυτές ε, διστάζουν να απευθυνθούν στην αγορά, ενώ υπάρχει πρόβλημα πιστώσεων σε πάρα πολλέ χώρες σήμερα, πολύ περισσότερο από ό,τι πριν από πέντε χρόνια. Άρα χρειάζεται χρηματοδότηση από διάφανες αγορές. Πρέπει να υπάρχουν πλατφόρμες με διαφάνεια που να επιτρέπουν τις συναλλαγές επενδυτή ε, και αποταμιευτή και να υπάρχει πλήρης διαφάνεια στις αγορές έτσι ώστε να έχουμε μια πραγματική οικονομία των αγορών. Αλλιώς θα έχουμε και έχουμε μη αγορά κερδοσκοπίας. Τώρα, για να έρθω στα πιο τεχνικά στοιχεία, θέλω να επιμείνω σε μερικά πράγματα που θα τα βρείτε έτσι κι αλλιώς στο γραπτό μου κείμενο. Έρχομαι πρώτα στην εμπορία των ε, οικονομικών προϊόντων. Υπάρχουν τρία στοιχεία κλειδί στις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το πρώτο είναι η απαγόρευση που προτείνεται ορισμένων προϊόντων, πρακτικών ή επικίνδυνων υπηρεσιών. Ε, θετικό αυτό διότι η καινοτομία δεν πρέπει να γίνεται σε βάρος της προστασίας των επενδυτών. Δεύτερον, εμπορία των περίπλοκων προϊόντων, όπως είναι τα ΟΣΕΚΑ, Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες. Εδώ μπορεί να υπάρξει βελτίωση για όλους τους ΟΣΕΚΑ μέσω στρατηγικών εναλλακτικής διαχείρισης. Και αυτό είναι κάτι το οποίο ε, πρέπει να φροντίσουμε ακόμα και όταν δεν προβλέπονται πράγματα στην παρουσίασή τους. Τρίτο θέμα είναι μια εγκάρσια πρωτοβουλία σε θέματα ενημέρωσης και προστασίας των επενδυτών, όποιο και αν είναι το προϊόν, είτε είναι τραπεζικό, είτε είναι ασφάλεια, είτε είναι παραγωγή. Η Επιτροπή προτιμάει μία κατά τμήματα προσέγγιση δηλαδή άλλα για τις τράπεζες, άλλα για τις ασφάλειες κλπ. Ενώ εμείς πιστεύουμε ότι δεν είναι αυτή η σωστή λύση. Γιατί ο σύμβουλος ή ο πελάτης έτσι δεν έχουν ενιαίο νομικό πλαίσιο. Δεύτερον τώρα, έρχομαι στην οργάνωση των αγορών. Εδώ χρειαζόμαστε ασφαλείς αγορές με διαφάνεια, προκειμένου να διασφαλίσουμε την ακαιρότητα των αγορών πρέπει ο ρυθμιστής να μπορεί να έχει πρόσβαση στις εντολές όλων των ε, πλατφόρμων, όλων των τόπων διαπραγμάτευσης όπου γίνονται συναλλαγές τίτλων. Το σύνολο των τόπων αυτών πρέπει να έχει την υποχρέωση εποπτείας των συναλλαγών που λαμβάνουν χώρα. Και εννοείται ότι πρέπει, όπως υπογραμμίστηκε ήδη, για να διασφαλιστεί η σταθερότητα των αγορών, να πάρουμε μαθήματα από το flash crash που έλαβε χώρα στην Wall Street και να φροντίσουμε να έχουμε ε, προβλέψει ένα πανευρωπαϊκό πλαίσιο έτσι ώστε η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών να μπορεί να ε, παρεμβαίνει. Πρέπει επίσης διαπραγματεύσεις να γίνονται μέσω μεταξύ πραγματικών αγορών, ε, δηλαδή των οργανωμένων αγορών ή του MTF. Η νέα πλατφόρμα πάντως, OTF, Μηχανισμός Οργανωσμένων Διαπραγματεύσεων, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στο στόχο αυτόν. Πρέπει να γίνει πιο φιλόδοξος και οι διαπραγματεύσεις να γίνονται σε πολυμερείς μηχανισμούς διαπραγματεύσεων, σε τέτοιες μόνο πλατφόρμες. Τέλος, πρέπει να προτείνουμε Πρώτα απ' όλα, οι συναλλαγές να καταγράφονται έτσι ώστε να μπορούν οι υποπτικές αρχές να βλέπουν ποιες είναι αυτές που δεν πρέπει να είναι αδιαφανείς. Δεύτερον, πρέπει να ε, βάλουμε περισσότερο φως στις ε, συναλλαγές που γίνονται εξωχρηματιστηριακά και τέλος πρέπει να φροντίσουμε περισσότερο για την προστασία των ε, επενδυτών. Ευχαριστώ. Ε, Μειώνοντα τις εξαιρεσει και τις αποκλήσει. Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε την κυρία Καόπη, την οποία θέλουμε να ακολουθήσουμε ως ε, Διευθύνοντα Σύμβουλα ε, της Ομοσπονδία Οικονομικών Υπηρεσιών της Φιλανδία. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους, ειδικότερα τον εισηγητή και τους κοιόδης εισηγητές που με καλέσατε ξανά στο Κοινοβούλιο. Είναι η πρώτη φορά που βρίσκομαι σε αυτή την πλευρά και με πολύ ενδιαφέρον ακούω όλα τα σχόλια για τη ΜΥΦΙΔ 1 ως εισηγητρία της ΜΥΦΙΔ 1. Χαίρομαι που κάναμε κάτι καλό με αυτή την νομοθεσία τελικά. Και τώρα περνάμε στην αναθεώρηση της ΜΥΦΙΔ που σίγουρα όπως είπε ο εισηγητής αποτελεί ένα από τους θεμελιώδεις λήθους ε, της ρύθμισης των κεφαλαίων αγορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πολύ σημαντική η συζήτηση που έχουμε σήμερα και είναι μεγάλη μου τιμή που βρίσκομαι εδώ μερικές παρατηρήσεις για την προστασία των επενδυτών. Οι προτάσεις βελτιώνουν την κατάσταση σε σχέση με τις προηγούμενες εκδόσεις. Υπάρχουν πολλές βελτιώσεις στην πρόταση της Κομισιόν σε σχέση με τη διαβούλευση, αλλά έχουμε ακόμη κάποιες, ε, κάποιους ενδιασμούς. Φυσικά υπάρχουν καθαροί κανόνες προστασία των επενδυτών με ίσους όρους ανταγωνισμούς, ανταγωνισμού, αγορές, και οι επενδυτές και οι καταναλωτές είναι σημαντικά θέματα για εμάς. Απομένουν μερικές πρότασεις όπου η επιχειρηματολογία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν μας πείθει. Αυτές οι προτάσεις περιορίζουν τις επιλογές δυσανάλογα. Υπάρχουν νέοι περιορισμοί και νέες ευθύνες που δεν αιτιολογούνται και που δεν βελτιώνουν ε, τους Ευρωπαίους τελικούς επενδυτές. Ε, μία από τις προκλήσεις είναι ότι δεν έχει περάσει αρκετός καιρός ε, ώστε να δούμε ποια ήταν ε, τα ωφέλη από την πρώτη MIFID ή να ανοιχνεύσουμε τα προβλήματα. Πίστευω ότι για παράδειγμα αυτές οι νέες επιτροπές καινοτομίε που δημιούργησε το Κοινοβούλιο και που καθιερώθηκαν λόγω του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα μπορούσαν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στο μέλλον όσον αφορά την υλοποίηση της ΜΥΦΙΤ 2. Επίσης, θα μπορούσαν να αποδειχθούν πολύ σημαντικές σε αυτή τη συζήτηση για το ποια προϊόντα είναι πολύπλοκα και ποια μη πολύπλοκα και για το ποιος θα πρέπει να είναι η προστασία των καταναλωτών εκ των, υστέρων, εκ προτέρων. Έχουμε συζητήσει ήδη για τις καινοτομίε και για... ήθελα να απαντήσω στα ερωτήματα του κ. Φέρμπερ. Χρειάζεται να συζητήσουμε αυτές τις απαγορεύσεις προϊόντων εξάντε. Οι χρηματιστηριακές εταιρείες που παρέχουν χρηματιστηριακές υπηρεσίες ε, είναι ικανές να παρέχουν επαρκή αξιολόγηση ε, των προϊόντων και του κατά πόσο αυτά αποτελούν απειλές. Είναι αυταποδεικτό ότι οι χρηματομεσίτες οι ίδιοι θα πρέπει να έχουν την ευθύνη να διασφαλίζουν ότι υπάρχουν οι σωστές διαδικασίες ε, κατά την ε, διαδικασία καινοτόμων προϊόντων η Εθνική Ρυθμιστική Αρχή θα πρέπει να μπορεί να παρεμβαίνει στη διαδικασία και να απαγορεύει ορισμένα προϊόντα από τη διάθεση στην αγορά. Ενισχύει την αντίληψη ότι υπάρχει γενική τάση των εθνικών ρυθμιστικών αρχών να προσθέσουν απαιτήσει σε αυτέ τι MIFID. Επίση πρέπει να θυμόμαστε ότι υπάρχουν τεστ καταλληλότητα για όλα τα πολυπλοκά προϊόντα, το οποίο αποτελεί πρόσθετη εγγύηση ότι δεν θα αποτελούν απειλή για συγκεκριμένου επενδυτέ. Για ποιο λόγο λοιπόν να απαγορεύσουμε τα πολύπλοκα προϊόντα ή τα διαρθρωμένα προϊόντα εκ των προτέρων. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Ειδικότερα επειδή έχουμε αυτές τις νέες επιτροπές για τις καινοτομίες αυτές μπορεί να παίξουν σημαντικό ρόλο στη διαδικασία και να εξετάζουν τις πρακτικές αγοράς επικεντρωμένες στην ενιαία αγορά και όχι κατά περίπτωση ανάλυση, κατά περίπτωση ανάλυση συγκεκριμένων προϊόντων. Το δεύτερο μου ζήτημα είναι η υπηρεσία μόνο εκτέλεσης. Ε, ρωτάει ο κύριος Φέρμπερ στο σημείο 16 πώς μπορούμε να καθορίσουμε τα πολύπλοκα και ποια είναι μη πολύπλοκα προϊόντα. Στο άρθρο 25 της πρότασης ε, η Κομισιόν αναφερόμενη στους κανόνες ε, εκτέλεσης δεν είναι σαφή. Θα χρειαστεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο να ζητήσει σωστή αιτιολόγηση. Η υπηρεσία μόνο εκτέλεση για μη πολύπλοκα προϊόντα είναι σημαντική για όλη τη χρηματοοικονομική βιομηχανία, για όλο το χρηματοοικονομικό τομέα και θα πρέπει να διατηρηθεί ω έχει όλε. Ε, οι τράπεζε των βόρειων χωρών χρησιμοποιούν ε, ε, αποδοτικές υπηρεσίες μέσω ίντερνετ. Δεν έχουν υπάρξει προβλήματα στις αγορές όσον αφορά αυτή την υπηρεσία. Γι' αυτό τον λόγο θεωρούμε ότι δεν υπάρχει λόγος για τις πιο αυστηρές ε, τροποποιήσεις που προτείνονται. Η νομοθεσία δεν μπορεί να απαγορεύει στους πελάτες να αγοράζουν επενδυτικές συμβουλές. Δεν μπορεί να ρυθμίζουμε τη συμπεριφορά των επενδυτών, αλλά να προστατεύουμε όσους ζητούν συμβουλές ή αξιολόγηση καταλληλότητας. Πρέπει να θυμόμαστε ότι οι υπηρεσίε εκτέλεσης χρησιμοποιούνται μόνο εφόσον τη ζητήσει ο πελάτης και ο πελάτη μπορεί να ζητήσει τεστ καταλληλότητας εφόσον χρειαστεί. Το να χωρίζουμε του χρήστε σε δύο διαφορετικέ κατηγορίε δεν έχει νόημα. Ο πελάτη θα πρέπει να μπορεί να χρησιμοποιεί υπηρεσίε μόνο εκτέλεση βάσει του άρθρου 25 τη MIFID. Πρέπει να θυμόμαστε ότι η πολυπλοκότητα δεν σημαίνει απαραίτητα κίνδυνο. Μπορεί να υπάρχουν πολύ πολύπλοκα προϊόντα που είναι λιγότερο επικίνδυνα για του τελικού επενδυτέ. Επίση, δεν υποστηρίζουμε την τροποποίηση με την οποία θα απαγορευτεί επιτευχθεί ο συνδυασμός της πίστοσης με μονοεκτέλεση. Το γεγονός της χρήσης αυτής πίστοσης δεν κάνει την συναλλαγή πιο περίπλοκη. Κάτι τέτοιο θα περιοριζει την υπηρεσία που παρέχεται από έναν πάροχο υπηρεσιας αλλά όχι την υπηρεσία που παρέχεται από ένα τρίτο μέρος Δεν έχει νόημα λοιπόν. Και τέλος, όσον αφορά την χρηματοοικονομικό τομέα, στην ερώτηση 15 ρώταει ο κ. Φέρμπερ αν υπάρχουν ανεξάρτητες συμβουλές ε, και κατά πόσο αυτό θα πρέπει να γίνεται χωρίς κίνητρα χρηματικά κίνητρα. Ο τρέχον κανονισμός είναι σχετικά νέος. Συνεπώς, πρώτα απ' όλα θα πρέπει να υλοποιηθεί σωστά αυτός ο κανονισμός και να αξιολογηθούν τα αποτελέσματά του. Προς το παρόν είναι πολύ νωρίς να αξιολογήσουμε τα πλέον τα αποτελέσματα αυτού του κανονισμού. Όσον αφορά τα κίνητρα έχουν περιγραφεί ε, πέρυσι σε κάποιο έγγραφο οι καλές και οι κακές πτυχές και αυτό το έγγραφο θα μπορούσε να λυθεί περισσότερο. Θα μπορούσαμε να το μελετήσουμε για να μελετήσουμε τα κίνητρα. Όσον αφορά τη διαχείριση χαρτοφυλακίου, συχνά τα κίνητρα ε, διαβιβάζονται τελικά στους ε, επενδυτές και δεν συμφέρει τους επενδυτές η απαγορευσή τους. Αυτό που ενδιαφέρει τους ε, πελάτες είναι το διασταυρούμενο κέρδος. Εάν το κέρδος δεν είναι επαρκές τότε ο πελάτης είναι δυσαρεστημένος και δεν θέλουμε πιο πολλούς δυσαρεστημένους πελάτες στην Ευρώπη. Συνήθω ο πελάτης εξετάζει το κόστος με τον ίδιο τρόπο. Εάν το κόστος και τα τέλη είναι ψηλά για ένα χαρτοφυλάκιο τότε είναι πιθανό αυτό το χαρτοφυλάκιο να εγκαταλειφθεί. η κατάργηση των κινήτρων θα οδηγούσε σε μείωση των υπηρεσιών που μπορούν να παρασχεθούν. Σε μια τέτοια περίπτωση θα μειωνόταν το εύρος των προϊόντων που προσφέρονται. Αλλά ουσιαστικά ε, ένα από τα πράγματα στο οποίο αποσκοπούσε η Μίφιντ είναι στο να υπάρχει ευρία επιλογή προϊόντων. Συνεπώς κάτι τέτοιο δεν θα ήταν ωφέλιμο για τους επενδυτές. Όσον αφορά τις ανεξάρτητες συμβουλές, η ορολογία στην πρόταση ΜΕΦΙΔ θα πρέπει να αλλάχθει. Όλες οι συμβουλές που παρέχονται από μεσίτες θα πρέπει να υφίσταται ένα τεστ καταλληλότητας και θα πρέπει να γίνεται προς το συμφέρον του πελάτη. Εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο θέλει να υποστηρίξει την πρόταση της Κομισιόν, Υπάρχει ένα συγκεκριμένο τύπο συμβουλών που παρέχεται από μια εταιρεία που εθελοντικά ισχυρίζεται ότι δεν λαμβάνει κίνητρα από τρίτο μέρο και συνεπώ οι συμβουλέ αμείβονται από τον πελάτη. Βάσει κάποιες αμοιβή. Συνεπώς δεν θα ήταν καλό να καταργηθούν αυτές, ή, ε, αυτά τα κίνητρα στις ιδιωτικές υπηρεσίες. Δεν έχουμε πιστικά, πιστήρια ότι η απαγόρευση λοιπόν η απαγόρευση λοιπόν είναι σωστά τεκμηριωμένη στην πρόταση της Κομισιόν. Χωρίς μικρόφωνο, κυρία Μακάρτη, δεν ακούγεται. Uh, ευχαριστώ. Δεν θα είμαι τώρα ελαστική ε, στο χρόνο σας. Κύριε Φέρμπερ, την ερώτησή σας. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Πολύ ενδιαφέρον το σημείο στο οποίο φτάσαμε και συναρπαστικό όταν ακούει κανεί τι τρει παρεμβάσει. Και έτσι, με την κυρία Ρο έχει κανεί την εντύπωση ότι εάν γίνει δεκτή η πρόταση της Επιτροπής ε, θα έχουμε ένα ευρύτατο περιθώριο απαγόρευσης εκ των υστέρων ενώ ίσως θα έπρεπε να διερωτηθούμε αν το εκ των προτέρων ο έλεγχος εκ των προτέρων θα μπορούσε να είναι η λύση Δηλαδή, το ερώτημα που μας απασχολεί είναι πρέπει να επιτρέπονται τα πάντα και όταν αρχίσει να ε, καταραίει η αγορά, όταν κάτι πάει στραβά, τότε θα σκεφτούμε να απαγορεύσουμε εκ των υστέρων κάποιο προϊόν. Επίσης είπε η κυρία Ρος ότι και προς, ε, και, και προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή φυσικά ότι μπορεί να έχουμε την ευρύτερη δυνατή νομοθετική ρύθμιση και σε εθνικό και σε συντονισμένο ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά εκ των υστέρων. Αγαπητή Πιανόρα πήγαν ώρα και εσύ ήσουν ε, από αυτή τη μεριά του Κοινοβουλίου, ξέρεις πολύ καλά ότι είναι η λύση όχι μόνο εκ των υστέρων έλεγχος, αλλά και ο εκ των προτέρων. Έχουμε το χρόνο μας να το συζητήσουμε. Αλλά. Επίσης, ε, ανεξάρτητη η μη παροχή συμβουλών. Από μια πλευρά βέβαια θα πρέπει να επισημάνω ότι να μην είναι σωστή η ορολογία που επιλέγεται, αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω, ίσω βρούμε κάποιο διαφορετικό όρο για τη μη ανεξάρτητη παροχή συμβουλών. Και ίσως θα πρέπει να το κοιτάξουμε λίγο πιο προσεκτικά. Εάν αυτό θα ισχύει ανεξαρτήτως ή αν θα πρέπει να συνδεθεί σε κάποιο συγκεκριμένο προϊόν με το φαινόμενο δηλαδή των κινήτρων ή μη. Είναι δηλαδή πιο χρήσιμη ενδεχομένω η διάκριση μεταξύ των προϊόντων από την διάκριση μεταξύ της ανεξάρτησης, η μη παροχής συμβουλών. Και επίση μια τελευταία παρατήρηση δεν είναι ερωτηματολόγιο του κυρίου Φέρμπερ, το άκουσα αρκετέ φορέ να λέγεται. Είναι ερωτηματολόγιο τη Επιτροπή των Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων. Μαζί το ετοιμάσαμε. Ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρο. Κυρία Ρο, κυρία Κάουπη, κυρία Ρο, πρώτα για το εκ των υστέρων. Yes, thank Κύριε Άρος, ε, πρόεδρε, είναι λεπτή ισορροπία, ξέρω, για, τον, ε, για τη ρυθμιστική αρχή να ζητήσει μια εκ των προτέρων έγκριση μεμονωμένων προϊόντων. Ξέρω ότι ορισμένα κράτη-μέλη τακτικά το πράττουν αυτό, η Γαλλική Αρχή παραδείγματι, ε, ΕΜΕΘ, αλλά άλλες όχι. Εν πάση περιπτώσει ξέρω ότι η τάση αυτή τη στιγμή είναι να προσφέρονται περισσότερα μέσα παρέμβασης όσο το δυνατόν πιο νωρί σιγά σιγά όλο και πιο νωρί στην διαμόρφωση αλλά και τη διάθεση στην αγορά των προϊόντων. Και ξέρω ότι η εξέλιξη αυτή είναι πολύ σημαντική. Βέβαια το ερώτημα παραμένει ότι δεν είναι δυνατόν πάντοτε να προβλέψουμε εκ των προτέρων τι είδους προβλήματα μπορεί να προκύψουν. Για ορισμένα προϊόντα ενδεχομένως να είναι ορατή τι η πιθανολόγηση να χάσει κάποιο επενδυτή ανεξαρτήτω των εξελίξεων και ανεξαρτήτω και τη πορεία του ίδιου του προϊόντο. Δηλαδή, μπορεί να μην μπορέσει να κερδίσει ποτέ ο επενδυτή. Οπότε, ενδεχομένω να θέλει κανεί να, να έχει μια πιο προληπτική δράση, να προλάβει δηλαδή τι εξελίξει. Αλλά για άλλα προϊόντα, ίσω χρειάζεται να περιμένει κανεί να δει τι εξελίξει στην αγορά για να δει τι είδου επίπτωση μπορεί να φέρουν και αναλόγως να δράσει, αλλά πρέπει εκεί να μπορεί να δράσει ταχαίως ε, ε, για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα όπου εμφανίζονται αυτά. Κυρία Κάουπη. Η κυρία Ρώσ νομίζω ήταν ακριβώς ε, πολύ συγκεκριμένη στην απάντησή της. Είναι πολύ δύσκολο εκ των προτέρων να προβλεφθεί ποια προϊόντα... Δεν νομίζω ότι είναι αυτό, λέει η Πρόεδρος, αλλά εν πάση συνεχίστε. Ποια προϊόντα μπορεί να είναι επιβλαβή για την αγορά. Ναι, αλλά μας εξήγησε ότι είναι πολύ δύσκολο να προβλεφθεί ποια προϊόντα είναι πιο επιβλαβή ή περισσότερο ή λιγότερο επικίνδυνα για τον πελάτη. Μας περιπτώσει λοιπόν, ε, γι' αυτό θα πρέπει να γίνεται εκ των υστέρων ο έλεγχος. Και όταν μίλησα για τις εκ των προτέρων απαγορεύσεις, τις αναφέρω μόνο και μόνο επειδή υπάρχουν εθνικές μενα Ορισμένα κράτη-μέλη υπάρχουν τέτοιου είδου προβλέψεις, διατάξεις, πρόνοιες για την εκ των προτέρων έγκριση των προϊόντων και μετά τη διάθεσή του στον επενδυτή, με προβλήματα στη διαδικασία αυτή. Φέρει πέντε στη Δανία. Υπάρχει λεγότερη σήμανση με τρία διαφορετικά χρώματα, πράσινο, πορτοκανί και κόκκινο. Σήμανση η οποία εν τέλει απεδείχθηκε όχι ορθή και οδήγησε επενδύσεις με εμπιστοσύνη πλευρά του επενδυτή στη σήμανση γιατί θεωρήθηκε ότι το προϊόν δεν ήταν τόσο επικίνδυνο, πράγμα όμω το οποίο επιδείχθη εισφαλμένη εκτίμηση. Και αυτό μπορεί να είναι νομίζω ένα στοιχείο στην αιτιολόγηση του ΜΜΕΦΙΔ, ότι υπάρχει αυτή η εμπειρία, υπάρχουν, έχουν γίνει σχετικέ ε, επαληθεύσεις και δεν μπορούμε να προβλέψουμε πάντοτε ένα, την πορεία ενός προϊόντος εκ των προτέρων. Από το, ε, το 1 με όλα τα κίνητρα που, για τα οποία θα πρέπει να ενημερώσουμε τον πελάτη, τον ε, επενδυτή κτλ. Ε, πάλι τώρα επανέρχεται το ζήτημα πως θα πρέπει να τα απαγορεύσουμε αυτά όλο, όλος διόλου. Αλλά τελικά το αποτέλεσμα είναι ότι ο πελάτης μάλλον βρίσκεται σε χειρότερη περίπτωση γιατί απευθύνεται στον ε, καταναλωτή, στον επενδυτή δηλαδή το κίνητρο. Επομένω, αν πρόκειται να δοθεί κάποια συμβουλή σε σχέση με κίνητρα στον καταναλωτή, στον επενδυτή, αυτή θα πρέπει η συμβουλή να δίνεται ανεξάρτητα, να γνωρίζουμε ότι είναι ανεξάρτητη ουδέτερη δηλαδή, βέβαια με το σχετικό αντίτιμο. Και σε μια διαφορετική κατάσταση όπου τα πράγματα είναι πολύ πιο δύσκολα, τότε δεν μπορεί να δοθεί κίνητρο, δεν μπορεί να δοθεί κίνητρο ούτε καν στη διαχείριση του χαρτοφυλακίου, αλλά τότε θα πρέπει να γίνει και η σχετική ενημέρωση, γιατί δεν μπορεί να υπάρχει αυτό με, το σχετικό, με τη σχετική επαλήθευση κινδύνου. Καλώ λέει ο πρόεδρο, να ακούσουμε τι ερωτήσει. Κύριε Γκέμπελ, έχετε κάτι, όχι. Να ακούσω του άλλου σκιώδει, τότε ο κύριο Σμιτ. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Θα ε, ήθελα να ρωτήσω την κυρία Τι είδου δυνατότητε μπορεί να έχουν οι αρχές και υποχρέωση για υλοποίηση των υποχρεώσεων που επομίζονται. Ξέρετε ότι εμείς από πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αγωνιζόμαστε πολύ για ενουσιαστικό έλεγχο. Θεωρείτε όμως ότι έχουμε τα, τα δημοσιονομικά μέσα το ανθρώπινο δυναμικό αλλά και τους ε, υλικοτεχνικούς πόρους ε, πληροφορικής κυρίως για να υλοποιηθούν όλοι αυτοί οι στόχοι και οι υποχρεώσεις. Και στο κρίσιμο ερώτημα περί κακών συμβουλών και απαγόρευσης. Εγώ, Πρόεδρε, το, την Άνοιξη ε, αγόρασα μετοχές της Τράπεζας Ιρλανδίας την Άνοιξη. Έχω χάσει ήδη 75%. Τι θα πρέπει να κλείσει η σχετική μονάδα στην τράπεζα της Σουηδίας. Όχι, δεν αστείευομαι. Γιατί είναι πολύ εύστοχο το ερώτημα της Πιανόρα. Είναι πολύ περίπλοκο το θέμα της ευθύνη την οποία αναλαμβάνει ο ίδιος ο πελάτης σε τελευταία ανάλυση. Και δεν πρέπει να δώσουμε την, δεν πρέπει να δώσουμε την εντύπωση ότι αυτού του τύπου οι επενδύσεις είναι απαλλαγμένες κινδύνου, γιατί δεν αποβαίνει σε όφελος του πελάτη, του καταναλωτή αυτό, του μικρού δηλαδή επενδυτή. Και συμφωνώ απολύτως ότι χρειαζόμαστε η καλύτερη νομοθεσία, πιο αυστηρή νομοθεσία, αλλά με πολύ μεγάλη σύνεση πρέπει να τη διαμορφώσουμε και πολύ ισορροπημένα. κυρία Κουίνπουρ, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Και ευχαριστώ την κυρία Ρος για τα σχόλιά της τα σχετικά με τα κίνητρα και το είναι ε, μεταχείριση των ανεξάρτητων ε, συμβουλών σε αντιπαράθεση με τις λοιπές λοιπού τύπου συμβουλές. Πρέπει να είμαστε πολύ σαφεί σε αυτό γιατί δεν υπάρχει άτομο πεδίο ανταγωνισμού και ταυτόχρονα το ζήτημα των επενδυτών από τρίτε χώρε. έτσι ώστε πάλι να έχουμε ανοιχτό περιθώριο για επενδύσεις ε, σε άλλες αγορές, άλλα προϊόντα. Έστω. Αλλά θα επικεντρωθώ εγώ σε δύο τομείς που δεν έχουν καλυφθεί. Οι αγορές ε, χονδρικής διαφοροποιούνται πολύ σχέση με τις μικρές αγορές, μικρές επενδύσεις. Δεν θα έπρεπε να έχουμε για τις μεγάλες αγορές χονδρικής του ΣΥΠΗΝ διαφορετικούς κανόνες και αντίστοιχα να λάβουμε υπόψη και επιχειρήματα που θα είχαν να κάνουν ε, στην περίπτωση των μικρότερων αγορών της Λιανικής με την αποτελεσματικότητα της ε, αγοράς. Για δε τα εξωχρηματιστηριακά δεν θα έπρεπε ενδεχομένω να κοιτάξουμε το επιχείρημα που θα οδηγούσε στο συμπέρασμα ότι εάν μειωθούν τα OTC τότε βελτιώνεται, ε, βελτιώνονται οι συνθήκες προστασίας του καταναλωτή, του επενδυτή. Ευχαριστώ κύριο Σκλουτέ. Ε, έχω μάλλον σχόλιο παρά ερώτηση. Αν κοιτάξουμε πόσο περίπλοκο είναι όλος αυτός ο χώρος και βέβαια και ο κύριος Σμιτ μας είπε ότι έχασε από μια επένδυση του αντίστοιχα μεγάλα ποσά. Ε, ερωτώ λοιπόν, είναι δυνατόν να εξασφαλιστεί μια αποτελεσματική προσφυγή του καταναλωτή και αν ναι, Το είπατε και εσείς κυρία Ρώσο ότι υπάρχει προστασία του επενδυτή, αυτή είναι η μία, η μία οπτική. Η άλλη οπτική είναι να εξασφαλίσουμε έναν τρόπο ορθολογικό αλλά και διαφανή για ενημέρωση του ενδιαφερομένου ε, που βεβαίως αποτελεί και προϋπόθεση της προστασίας του καταναλωτή. Αλλά πώς μπορούμε να του εξηγήσουμε τον κίνδυνο και να τον καταστήσουμε αντιληπτό, κατανοητό τον κίνδυνο αυτόν και απτό για τον ίδιο τον καταναλωτή. Ευχαριστώ κύριο Γκοζέ. Όχι, λάθο έκανα. Χωρί μικρόφωνο. Καλό. σα απαντήσει ο κύριο Βουέι πρώτα, παρακαλώ, μια και ήταν ο τελευταίο που μίλησε νωρίτερα. Σα ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μου δίνετε το λόγο και την κυρία Ρώση που μου παραχωρεί τη θέση της. Είναι πολλοί οι λόγοι για του οποίους ε, λυπούμε που δεν έχω γίνει ευρωβουλευτή, Πάντοτε απολαμβάνω ιδιαίτερα όποια συμμετοχή έχω εδώ στο Κοινοβούλιο και λυπούμε που δεν έχω και την ίδια ε, ευγλωτία και ευχέρεια λόγω με την κυρία Κάουπη που βέβαια έχει θητεύσει εδώ. Αλλά για να είμαι λίγο πιο σοβαρός. Όχι, όχι. Ξέρει πολύ καλύτερα από ότι εγώ πώς να χειριστεί τον λόγο και πώς να αξιοποιήσει το χρονικό περιθώριο που της δίνεται. Εν πάση περιπτώσει όμως, πιο σοβαρά τώρα, θα ήθελα να πω στον κύριο Φέρμπερ, που συμφωνώ απολύτως μαζί του, ότι πιο σημαντικό από το να δούμε αν έχουμε ανεξάρτητες ή συμβουλές, είναι να έχουμε διαφάνεια και διαδικασία για ε, ρύθμιση συγκρούσεων συμφερόντων. Αυτό είναι νομίζω το πιο σημαντικό για την προσοχή του επενδυτή. Και δεύτερον, στην ε, Γαλλία και του υπογράμμιση Έχουμε παράδοση εκ των προτέρων με όλη την περιπλοκότητά τους να ελέγχουμε τα προϊόντα, τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα και δεν υπάρχει κανένας λόγος όπως ρωτήθηκε νωρίτερα να περιοριστούμε σε μια ρύθμιση η οποία θα επέτρεπε μόνο εκ των υστέρων έλεγχο. Όχι, στη Γαλλία μπορούμε εκ των προτέρων να ελέγχουμε, όχι οφείλουμε να ελέγχουμε εκ των προτέρων τα προϊόντα και δεν βλέπω ότι θα πρέπει να περιοριστούμε μόνο σε μια εκ των υστέρων ε, παρακολούθηση, έλεγχο κτλ. Οφείλουμε να κάνουμε λοιπόν τον, τον εξάντα έλεγχο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν έχουμε δυναμική στις αγορές μας και άλλωστε έχουν πολλά προϊόντα επιβιώσει κατά αυτόν τον τρόπο και άλλωστε αναφέρθηκα. Και τώρα η Βερένα για να μιλήσει για τις πραγματικές εξουσίες. Για να απαντήσω σε κάποια από τα ερωτήματα που ακούστηκαν νωρίτερα πριν επανέλθω στις ανεξάρτητες συμβουλές. Είναι πιστεύω σημαντικό, όπως είπε και ο Ζομπιέρ, να είναι σαφές το ποιος δρά, με ποια ιδιότητα συμβούλου και γιατί είναι στο συμφέρον δρά. Και έτσι τουλάχιστον ο πελάτη δεν πέφτει θύμα συγκρούσεων συμφερόντων από κάποιο σύμβουλο με σκοτεινά συμφέροντα ή μη ε, ομολογημένες σχέσεις. Αυτό νομίζω απαντά και στον κύριο Σμιτ. Ναι, έχει ο πελάτη ευθύνη ο ίδιο. Ισχύει το κάβε attemptor, δηλαδή ο αγοραστή πρέπει να γνωρίζει τι κάνει, έχει την εφέρει την ευθύνη τη αγορά του. Αλλά παρόλα αυτά θα πρέπει να είναι σε θέση και να εμπιστεύεται τη συμβουλή που του χορηγείται. Και, εν πάση περιπτώσει, αν κανείς ασχολείται με ένα προϊόν μόνο επί τη βάση τη εκτέλεση, ξέρει ότι, είναι, ότι αναλαμβάνει ο ίδιο τον κίνδυνο. Εάν όμω ε, πιστεύετε έναν σύμβουλο, αν λαμβάνει συμβουλέ από κάποιον ειδικό, τότε θα πρέπει να μπορεί και να τον εμπιστευτεί. Για τις αγορές ε, ομολόγων και λιανικής ε, ή χονδρικής και βέβαια εξωχρηματιστηριακών χρηματιστηριακών ε, ε, μέσων. Βεβαίω μπορούν να γίνουν διακρίσει, υπάρχουν διαφορετικά μεγέθη στι συναλλαγέ, επισημάνθηκαν ήδη, υπάρχουν διαφορετικοί τύποι αγορών, και δεν μπορούμε να πούμε ότι μπορεί μία προϋπόθεση που ισχύει για την αγορά των μετοχών να ισχύει 100% σε κάθε άλλο τύπο και μέγεθος αγοράς. Βεβαίως χρειάζεται περισσότερη διαφάνεια εν γέννη όμως ε, σε όλες ε, τις αγορές ε, και πιστεύω ότι αυτό ισχύει και για την αγορά των ομολόγων εν γέννη, για τις αγορές των ομολόγων, για τα εξωχρηματιστηριακά, τα OTC η μείωση συναλλαγές αυτών ε, θα βελτιώσει, λέτε, την ε, προστασία του καταναλωτή. Εν πάση περιπτώσει, η απάντηση μου είναι ότι θα βελτιώσει τις συνθήκες διαφάνειας στην αγορά. Και άρα αυτό πιστεύουμε ότι εν τέλει τίνει προς την βελτίωση της προστασίας του καταναλωτή. Του επενδυτή δηλαδή. Αλλά θα πρέπει να κοιτάξουμε βέβαια και άλλα μέτρα που άλλωστε εξετάζει και η πρόταση MIFID ε, με στόχο βέβαια να γίνουν πιο διαφανείς οι αγορές για τον επενδυτή, το μικρό επενδυτή. Καλώ λέει η Πρόεδρο και για να ε, η κυρία Ρώσ, και για να επανέλθω στην ερώτηση του κυρίου Σμιτ για τι ε, προκλήσει τη ΜΥΦΙΤ. Με χαρά βλέπω ότι επιτρέπεται μέσω αυτή ένα νέο δημοσιονομικό κανονισμό που θα οδηγήσουν ουσιαστική τη υλοποίηση εν τέλει αλλά βέβαια αυτό θα είναι και η μεγάλη πρόκληση των προσεχών ετών. Ήδη επεξεργαζόμαστε την ΟΗΦΙΤΜΕΝ, τα αποτελέσματα όμως θα τα δούμε όταν τεθεί ουσιαστικά σε εφαρμογή αυτή. Είναι μεγάλη πρόκληση για μας. Και αναφερθήκατε Φερρυπίν στα θέματα της ε, τεχνολογίας, ε, της πληροφορικής. Το να σχεδιαστεί ένα ε, σύστημα πληροφορητικής για τον τελικό χρήστη, δηλαδή τον επενδυτή, ώστε να μπορεί αυτός να παρακολουθεί την αγορά, την λειτουργία της αγοράς, θα είναι τελικά η μεγαλύτερη δυσκολία. Κυρία Κάουπη. Ευχαριστώ για τα ότι και τι είναι υπέρ της προστασίας του επενδυτή. Λέω το ίδιο αυτό που είπα και στην αρχή στις παρατηρήσεις μου, ότι ο πελάτης επενδυτής θέλει ε, διασταυρούμενα κέρδη και οι ρυθμίσεις όντως έχουν μειώσει το κόστος συναλλαγής. Αλλά αυτό που ρωτήσατε κι εσείς για τις post-trade ε, υποδομές που δεν έχουν μειωθεί εξίσου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όντως έκανε κάποια λάθη σε αυτό το τομέα. Εμείς για χρόνια βασιστήκαμε στους κώδικες διοντολογίες και σε διάφορους ήπιους μη δεσμευτικούς κανόνες πράγμα που είχε σαν αποτέλεσμα να μην εξελίχθηκε πολύ η κατάσταση όσον αφορά αυτό το κόστος. Αλλά έχουμε προτάσεις από την Επιτροπή πιο σημαντικές σε αυτό το τομέα από ότι οποιασδήποτε άλλες αξίες συναλλαγών. Τώρα για τους οικονομικούς ε, πόρους. Είναι πολύ σημαντικό για τους ΣΕΚΑ να έχουν αρκετούς πόρους, να έχουν αρκετό προσωπικό και είναι προς το συμφέρον των Ευρωπαίων καταναλωτών και των πελατών γενικότερα να λειτουργεί καλά ε, να λειτουργούν καλά οι επενδύσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να φροντίσει να υπάρχουν όντω αρκετοί πόροι για αυτή την τόσο σημαντική λειτουργία. Κύριε Κοζέ, τώρα έχετε μια ερώτηση. Ναι. Αφήνω τον Μάρκο να ασχοληθεί με τα τεχνικά. Αλλά εγώ θέλω να αναφερθώ λιγάκι στα μέσα που έχουν οι διάφορες αρχές, η ΕΣΜΑ κλπ. Οι αρχές αυτές, η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών δηλαδή και Αγορών κλπ. είναι πραγματικές εξουσίες. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί πώς οργανώνονται και πώς χρηματοδοτούνται και πώς αποκτούν προσωπικό. Και επιμένω, γιατί εδώ βλέπουμε τη σχιζοφρένεια των κρατών, βλέπουμε ότι είναι χάρη στο Κοινοβούλιο που τελικά δόθηκαν οι αναγκαίες πιστώσεις, αυτές δηλαδή που προτάθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μπόρεσαν να αποκατασταθούν στον προπολισμό του 2012, ενώ τα κράτη-μέλη τι θέλανε, θέλανε μείωση κατά 50% και για την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών και για άλλες. Με το Λαμασούρ όμως τα καταφέραμε να υπάρξουν οι κατάλληλες πιστώσεις, οι οποίες ελπίζουν να αυξηθούν στο μέλλον, γιατί είναι αναγκαίο οι τρεις ε, αρχές, οι επιπτικές, να παίζουν ένα σημαντικό ρόλο όσον αφορά τις οικονομικές υπηρεσίες, τις τράπεζες και τις ασφάλειες. Ευχαριστούμε κύριε Κωσές. Κάτι κάνουμε καλό. Μερικές φορές κάνουμε λάθη, αλλά αυτό το πετύχαμε τουλάχιστον. Κύριε Φέρμπερ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Μια σύντομη παρατήρηση μόνο. Αλλά έφυγε ο κύριο Σμιτ. Εγώ μπορώ να πω ότι βλέπω ένα παραλληλισμό μεταξύ αυτής της νομοθεσίας και της νομοθεσίας για τα τρόφιμα. Ε, δηλαδή επιτρέπεται να κυκλοφορεί ένα προϊόν εφόσον επιβεβαιώνεται ότι δεν είναι επικίνδυνο. Στην περίπτωσή μου σοκολατάκια Βελγίου. Ε, και γι' αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να επιτρέψουμε να υπάρχουν τα προϊόντα τεχματοπιστωτικά εφόσον πάλι δεν είναι επικίνδυνα, εφόσον μπορούν να λειτουργήσουν σωστά. Χωρίς να υπάρχει πάντα η εγγύηση ότι δεν ενέχουν κανένα κίνδυνο, αλλά τουλάχιστον να μην περιλαμβάνουν συστημική διακινδύνευση. Αυτό είναι που αντιμετωπίσαμε σαν πρόβλημα στο παρελθόν, που δεν μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε στο παρελθόν. Και γι' αυτό τίθεται για μένα το ερώτημα. Στην πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αυτή η ΕΚΑ έχει περιθώριο να επιβάλλει απαγορεύσεις γενικές ουσιαστικά. Δηλαδή να απαγορεύσει τα πάντα μέσα από μια διάταξή της. Εκ των υστέρων αλλά δεν προβλέπεται τίποτα εκ των προτέρων, πράγμα το οποίο μου φαίνεται σαν να έχουμε μια άνηση κατανομή των ε, μέσων αντιμετώπιση των προβλημάτων. Και νομίζω ότι αυτό θα μα απασχολεί στου επόμενου μήνε. Με αυτό θα σπαζοκεφαλιάζουμε. Στο να εξασφαλίσουμε μια καλή ισορροπία. Αλλά και πάλι, όπω είπα, βλέπω ε, παραλληλισμό και σε αυτό, στη δυσκολία δηλαδή τη διαδικασία, τον παραλληλισμό με την ε, νομοθεσία περί τροφίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βεβαίω και υπάρχει απαγόρευση εκ των υστερών, αλλά υπάρχει και η εκ των προτέρων αδειοδότηση, σήμανση και το καθεξής. Και αυτό νομίζω είναι το χαρακτηριστικό, ότι βεβαίως ε, και θα πρέπει οτιδήποτε είναι δυνατόν και λογικό να επιτρέπεται, αλλά δεν θα πρέπει και να θεωρεί κανείς ότι οτιδήποτε επιτρέπεται είναι απαλλαγμένο παντό κινδύνου. Αυτά, αυτή είναι η λογική, το λογικό συμπέρασμα πιστεύω. Α απαντήσει η κυρία ρό Εκά για να επανέλθουμε. Πολύ σύντομα, ναι. Οι εξουσίες της ε, ΕΣΜΑ, της Ευρωπαϊκή Αρχής των Αξιών και Αγορών, είναι πολύ περιορισμένες. Έτσι συντονίζει τις εθνικές προσεγγίσεις και περιορίζεται από διάφορες διατάξεις ε, ότι δηλαδή πρέπει τα προϊόντα αυτά να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην ε, σταθερότητα τιμών, στην ευημερία κτλ. Δεν ε, πρόκειται δηλαδή για μια κάλυψη η Ευρωπαϊκή Αρχή Αξιών και Αγορών δεν μπορεί σε καθημερινή βάση να παρεμβαίνει για τα πάντα. ακόμα και αν μπορούσα να απαγορεύσω κάτι, ναι, είναι κάτι που προβλέπεται, αλλά δεν είναι κάτι που χρησιμοποιούμε σε καθημερινή βάση. Οι διατάξεις που προτείνει η Επιτροπή πάντως ε, ακριβώς διασφαλίζουν να πρόκειται για ένα συντονισμένο μηχανισμό με διάφορες ρήτρες ασφαλείας. Πρόεδρος, θα επανέλθουμε δίχως άλλο σε αυτό το θέμα και με τον εισηγητή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις εξαίρετες αυτές παρεμβάσεις σας και τις απαντήσεις σας. Θα συνεχίσουμε για περνάμε στο τρίτο τμήμα μας που αφορά την οργάνωση των αγορών και των διαπραγματεύσεων. Ξέρω ότι πολλοί ενδιαφέρονται για τις ε, νέες κατηγορίες των ε, τους μηχανισμούς δηλαδή οργανωμένων διαπραγματεύσεων, τι γίνεται με τα παράγωγα επί εμπορευμάτων, Όλα αυτά είναι πολύ ενδιαφέροντα και το πάνελ μας είναι πολύ σημαντικό επίσης και σας ευχαριστούμε που ήρθατε. Ο πρώτος είναι ο κύριος Τσερούτη, ο οποίος μας έδωσε μια γραπτή παρέμβαση και εκτενή που θα κυκλοφορήσει στους ευρωβουλευτές. Οπότε σας παρακαλώ να πάρετε το λόγο. Είσαστε πρόεδρος και αναπληρωτής εγκλησικός διευθυντής της είναι Euronext. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ και σας ευχαριστώ που με καλέσατε να έρθω εδώ σήμερα. Έρχομαι στο πρώτο ερώτημα όσον αφορά τις ε, υποχρώσεις και τις ρυθμίσεις στις πλατφόρμες διαπραγμάτευσης μεταξύ άλλων κατά πόσο περιλαμβάνεται και ο μηχανισμός οργανωμένων διαπραγματεύσεων και κατά πόσο τηρείται η αρχική νομοθεσία. Η MIFID 1 δημιούργησε περισσότερο ανταγωνισμό, επέτρεψε περισσότερες επιλογές, το έχουμε πει αυτό, υπάρχουν ε, νέοι που έχουν μπει στον ε, τομέα στις διαπραγματεύσεις και πρόκειται για ένας από τους νέους που, που έχουν μπει στην αγορά αυτή και έχουν μεγάλο μέρος της αγοράς είναι ο XC. Έτσι λοιπόν, GX. Έτσι λοιπόν, υπάρχουν στις πλατφόρμες κάτι που κυριαρχούν. Εμείς θέλουμε ένα ξεκάθαρο καθεστώς ε, για τις περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων σε συνδυασμό με τους κατόχους πλατφόρμας αλλά και με ε, τα κεφάλαια που κυκλοφορούν από τους πελάτες. Επίσης θέλουμε να υπάρχουν οι ίδιοι κανόνες στις ρυθμισμένες αγορές και ε, στις διαπραγματεύσεις του πολυμερή μηχανισμού. Ο κατακαιρματισμός με τις ε, ε, αγορές διαφάνειας, όπως είπαμε και πριν, έχει σαν αποτέλεσμα να είναι ο ρυθμιστής ο οποίος θα φροντίσει για την ισορροπία. Σήμερα δεν έχει επιτεθεί πλήρως η ισορροπία αυτή. Έχει υπάρξει μια ισορροπία ανάμεσα ε, στο, στη διαφάνεια. Εκεί υπάρχει κάποια ισορροπία. τεχνικά για τις διαπραγματεύσεις, όπως είπαμε ήδη, ένα μεγάλο μέρος των OTC, των over the counter δηλαδή, είναι στις ρυθμιζόμενες αγορές. Όσο πάντως δεν υπάρχει νομικός ορισμός, τότε οποιαδήποτε καινοτομία κινδυνεύει να οδηγήσει στις αδιαφανείς συναλλαγές. Γι' αυτό και λοιπόν πρέπει να καθορίσουμε τι είναι οι συναλλαγές οι εξωχρηματιστηριακές και να είναι πιο συγκεκριμένος ο ορισμός. Πρέπει με αυτόν τον τρόπο να διορθώσουμε ό,τι πάει στραβά σήμερα. Έρχομαι τώρα στα OTFs. Εμεί χαιρόμαστε για το γεγονό ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βλέπει ότι υπάρχει ένα πρόβλημα με τα παραθυράκια. Δεν πρέπει όμω να υπάρξει η δημιουργία περισσότερων κατηγοριών, γιατί νέοι τύποι πλατφόρμα ε, κινδυνεύουν να μπουν πάλι στην κατηγορία των έξω χρηματιστηριακών συναλλαγών. Η εισαγωγή τώρα μια τέταρτη κατηγορία θα έπρεπε να εξαρτάται από τον δεσμευτικό ορισμό των ε, εξωχρηματιστηριακών συναλλαγών. Για τα χαρακτηριστικά που προτείνονται για το OTF. Πρέπει να είναι εκτελεστές οι προδιαγραφές και προτείνεται να έχουν διακριτική ευχαίρεια όσον αφορά τις τιμές, αλλά αν οι τιμές δεν είναι δεσμευτικές, τότε η συνεισφορά τον OTF στη διαμόρφωση τιμών είναι κάτι που δεν έχει νόημα. Η πρόταση της Επιτροπής επίσης λέει ότι οι OTF δεν πρέπει να μπορούν οι ίδιοι να βάζουν δικά τους κεφάλαια, μια που και αυτοί όπως και οι αγορές δεν μπορούν να το κάνουν και μόνο μέσω του καθεστώτος ε, συστηματικής εσωτερικής να μπορεί να γίνει αυτό. Συνεχίζονται συζητήσεις για αυτό το θέμα σήμερα και πιστεύουμε ότι οι αλγοριθμικές διαπραγματεύσεις δεν είναι οι ίδιες όπως είναι η OTF. Υπάρχει μια διαφορά μεταξύ των δύο. Και ακριβώς πάνω σε αυτό είναι που συνεχίζει τη συζήτηση. Οι υψηλή συχνότητα ε, συναλλαγές είναι κάτι διαφορετικό από τις αλγοριθμικές. Δεν πιστεύουμε επίση ότι πρέπει να δαιμονοποιούνται από κάθε άποψη. Αναγνωρίζουμε ότι υπάρχουν μερικά προβλήματα που πρέπει να λυθούν για τι συναλλαγές αυτές, ε, ε, κατάχρηση στην αγορά, εντάξει δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία γι' αυτό. Το μέγεθός τους επίσης ως ποσοστό στην αγορά που είναι 70% και 32 50% στην ευρωπαϊκή αγορά μπορούν να δημιουργήσουν ε, ρευστότητα αυτό είναι συζητήσιμο. Έρχομαι τώρα στη δεύτερη ερώτηση που έχει να κάνει με τα παράγωγα επί εμπορευμάτων. Προτείνει κάποιες διατάξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που απορρέουν και από του ομάδα των 20. Εδώ όμω έρχονται οι ανησυχίε μα για την σταθερότητα των τιμών και για την μόχλευση που εξαρτάται από τις δυνατότητε παραγωγή. Υπάρχει ένα στοιχείο του προγράμματος δράσης που έχει να κάνει με την αγορά παράγωγων επί εμπορευμάτων. Υπάρχουν ε, δύο στοιχεία στην πρώτη επιτροπή που είναι μεγαλύτερη διαφάνεια και διαχείριση για σπόσα θέσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε ότι πρέπει να καθορίζεται θέση ανάλογα με την ε, κατάσταση του επενδυτή. Εμείς πιστεύουμε ότι κάτι τέτοιο θα βοηθήσει να ανακτηθεί πιστοσύνη στην αγορά. Η μόνη πρότασή μας για βελτίωση της πρότασης της Κομισιόν είναι να αφαιρεθεί η απαιτήση αναφοράς θέσης από τις εταιρείε μέλη σε πραγματικό χρόνο. Διότι η αναφορά σε πραγματικό χρόνο δεν αναφε... Ε, παράγει απαραίτητα μία σωστή έκθεση χρόνου, αλλά δημιουργεί πολλά προβλήματα. Τέλος, όσον αφορά τις ε, προτάσεις της Κομισιόν για τη διαχείριση θέσης, πιστεύουμε ότι ο αυστηρός έλεγχος στις αγορές παραγόγων είναι βασικό στοιχείο για τη διασφάλιση της σωστής λειτουργίας των αγορών. Η Κομισιόν έχει προτείνει οι τόποι διαπραγματεύσεων να επιβάλλουν όρια θέσεων με τα ίδια για την υποστήριξη της ρευστότητας, την πρόληψη της κατάχρησης της αγοράς και τη διασφάλιση των κανόνων. Υποστηρίζουμε αυτούς τους στόχους πολιτικής. Επίσης πιστεύουμε ότι η ύπαρξη εναλλακτικών διευθετήσεων με αντίστοιχα αποτελέσματα είναι βασικά διότι οι δομές των αγορών είναι πολύ διαφοροποιημένες και οι ρυθμιστικές λύσεις θα πρέπει να προσαρμοστούν σε αυτές. Τα όρια θέσεων για τις εναλλακτικές διευθετήσεις φυσικά θα πρέπει να εφαρμόζονται σε μια ευρύτερη διαδικασία διαχείρισης θέσεων. Τα όρια θέσεων μπορούν να αποτελέσουν χρήσιμη προσθήκη στις ε, ρυθμιστικούς κανόνες. Ε, η χρήση τους πρέπει να εξτοχευθεί προσεκτικά διότι τα όρια θέσεων μπορεί να διαστρεβλώσουν τις συνθήκες στην αγορά. Εάν εφαρμοστούν λανθασμένα μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα στη λειτουργία της αγοράς. Χρειάζεται διευκρίνηση για το κατά πόσο άλλες αρχές θα πρέπει να ε, επιβάλλουν κάποιες πρακτικές, όπως η Κομισιόν. Ολοκληρώνω λοιπόν εδώ. Well, I think we're going to leave that up to the competition authorities. That's not really for MIFID to regulate. Um, miss, the next person. Το επόμενο άτομο στη, λίστα μου είναι ο κύριο Σλούτερ. Παρακαλώ, έχετε τον λόγο. Ευχα... Κυρίες και κύριοι, συνάδελφοι, κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ θερμά για την ευκαιρία που μου δίνετε να σας ε, απευθύνω τον λόγο για την ε, νέα αυτή νομοθεσία MIFID που προτείνεται ως εκπρόσωπος του κλάδου. Και θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω, τις βιομηχανίες λένε, θα ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά τα προσεχή λεφτά για μένα. Έχουν τεράστια σημασία ακόμη και για την επιβίωσή μας. Και θα ήθελα, αν μου επιτρέπετε, να σας παρουσιάσω όλο τον, το προβληματισμό στον οποίο κινείται όλη η βιομηχανία. Με παράδειγμα τη δική μου την επιχείρηση, την Dream Aluminium Anonymous Εταιρεία διότι ως παραγωγός πρωτογενούς, δηλαδή πρώτης ε, τήξης αλουμινίου, με σχετικά χιτήρια, χώρους ανακύκλωσης και λοιπή ε, παραγωγή, ε, πληττόμαστε ιδιαίτερως από την προτινόμενη οδηγία. Δηλαδή είμαστε ένας χαρακτηριστικός εκπρόσωπος της πραγματικής οικονομίας. Εμείς ως προς το κόστος εξαρτώμαστε και από, για την αγορά των ε, πρώτων υλών μας, εξαρτώμαστε και από τον άργυλο και τα παλαιοσίδερα το, τις τιμές ε, του ηλεκτρικού ρεύματος του φυσικού αερίου αλλά και για την πώληση των προϊόντων μας εξαρτώμαστε από την πώληση του αλουμινίου και από τον κίνδυνο ισοτιμιακών, ε, ισοτιμιών μεταξύ ε, ευρώ και δολαρίου. Άρα λοιπόν δεν θα μπορούσαμε χωρίς τη δυνατότητα των μέσων διαφύλαξης προστασίας των, της αγοράς να επιβιώσουμε. Έχουμε να κάνουμε 500.000 τόνους προϊόντων αλουμινίου κάθε χρόνο για τους οποίους ε, χρειαζόμαστε 5 τεραβάτ ε, τεραβατόρες ηλεκτρική ενέργεια με κόστος σε, για το ηλεκτρικό ρεύμα 250 με 300 εκατομμυρίων ευρώ ανά χρόνο που επίσης ε, πρέπει να ασφαλίσουμε έναντι του κινδύνου. Ε, πρέπει να σημειώσω δύο ότι το ηλεκτρικό το πληρώνουμε σε ευρώ, αλλά τα προϊόντα μας τα πολλούμε σε δολάριο. Και άρα χρειάζεται να προστατευτούμε εναντί αυτών διακυμάνσεων και ταυτόχρονα να προστατεύσουμε και τον πελάτη μας εναντί της πτυτικότητας των τιμών. Το εμπόριο λοιπόν αυτό στο αλουμίνιο έχει να κάνει, ε, αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της πραγματικής ε, οικονομίας με ε, χρήση χρηματοπιστωτικών προϊόντων για την λειτουργία της, των οικονομικών κύκλων, χωρίς επίδραση όμως στο χρηματοπιστωτικό τομέα. Και έτσι αποδεικνύεται ότι δεν, μπορούμε να δεν αποτελούμε εμείς ποτέ ε, συστημικό κίνδυνο. Ωστόσο, κίνδυνοι επιμόλυνσης από την αγορά μέχρι στιγμής δεν υπήρξαν, ούτε και αναμένεται να υπάρξουν. Ε, αυτό αποδεικνύει άλλωστε η ιστορία μας από 130 χρόνια δραστηριοποίηση στο οργανωμένο τελικό εμπόριο με μη σιδηρούχα μεταλλεύματα. Εκτός ε, αυτών έχει αποδείξει η περίπτωση ένρων πριν από 10 χρόνια ότι ακόμη και μια μεγάλη ε, επιχείρηση ενέργειας δραστηριοποιούμενη σε παγκόσμιο επίπεδο μπορεί να ε, μην έχει κανένα κίνδυνο συστημικό για την μορφοπιστωτική αγορά. Εάν όμως επηρεαστούμε, αντιμετωπιστούμε κατά τρόπο ισότιμο με αυτό που αντιμετωπίζονται οι τράπεζε, τότε απλώ θα έχουμε αρκετά χρήματα και το χρήμα στη διάθεσή μα για να επιτελέσουμε το έργο μα, για να προβούμε στι συναλλαγές μα. Αυτό θα έχει τεράστιε συνέπειε και στο εργατικό μα δυναμικό και βέβαια σε ολόκληρο το ευρωπαϊκό επίπεδο στου πελάτε μα, δηλαδή τη βιομηχανία που αγοράζει τα προϊόντα μα όπω είναι αυτοκινητοβιομηχανία, η κατασκευαστική, ο κλάδο των εργαλειομηχανών, μηχανών κτλ και της συσκευασίας. Θα έχουμε πολύ χαμηλότερη ε, ρευστότητα στην αγορά και οι κίνδυνοι στην πραγματική οικονομία θα ε, σήμαιναν ταυτόχρονα και πολύ σημαντικές, σημαντικούς κλειδονισμούς στο σύστημα των τιμών. Πέραν αυτού, η συγκέντρωση στον χώρο των ε, ε, ενεργειακών και των πρώτων υλών μπορεί να θεωρηθεί ως δεδομένη εξέλιξη αν συμβεί κάτι τέτοιο. Σταθερή αγορά προφανώς χρειάζεται περισσότερες, από, περισσότερες επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε αυτήν, αλλά η οδηγία ε, MIFID δεν μπορεί να αντιμετωπίσει ε, το ζήτημα των OTC, των εξοχματιστριακών δηλαδή παραγόγων και δεν θα πρέπει να ε, επιδεινωθούν οι συνθήκες για τις επιχειρήσεις μη χρηματοπιστωτικού χαρακτήρα που ε, προβλέπεται να καλυφθούν τώρα από την ΜΥΦΙΤ. Επιτρέψτε μου λοιπόν να εξηγήσω και τι σημαίνουν τα όρια ως προς τις θέσεις, τα position limits. Για να έχουμε μια ουσιαστική αποτροπή κινδύνου θα πρέπει να ε, αγοράζουμε μακροπρόθεσμα ε, ε, ενέργεια και να πολλούμε μακροπρόθεσμα αλουμίνιο, πράγμα το οποίο συνεπάγεται αυτόματα υψηλές θέσεις. Με τα όρια, τα position limits δηλαδή, αυτή η δυνατότητα περιορίζεται σημαντικά για μας και όσοι εκ δεν θα μπορούμε ούτε να ασφαλιστούμε, δεν θα μπορούμε δηλαδή να δρούμε μόνο σε στενά όρια, σε στενά limits και άρα θα μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τη μεγάλη πτυτικότητα των αγορών ε, μετάλλων ούτε να αντιμετωπίσουμε τη πτυτικότητα ε, των τιμών της ενέργειας. Γι' αυτό λοιπόν παρακαλώ μην ε, επιτρέψετε αυτές τις ρυθμίσεις μόνο με μια πλήρη απελευθέρωση μπορείτε να προσφέρετε τη δυνατότητα και για μας αλλά και για ολόκληρη τη βιομηχανία σε 10 χρόνια να εξακολουθούμε να ε, λειτουργούμε ακόμη επικοδομητικά και αποτελεσματικά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω το λόγο στον τελευταίο μιλητή, στην κυρία Ζίζελ Ενρίκες από την ε, Διεθνή Συμμαχία Καθολικών Αναπτυξιακών Υπηρεσιών. Ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε την ευκαιρία να μιλήσω σε αυτή τη σημαντική ακρόαση με μέρου κοινων... της κοινωνίας των πολιτών και των οργανισμών της που ανησυχούν για τις επιπτώσεις της χρηματιστικοποίηση των τροφίμων. Τα παράγωγα που βασίζονται στα προϊόντα τροφίμων θέτουν σε κίνδυνο την επιστημιστική ασφάλεια εκατομμυρίων ανθρώπων. Για πρώτη φορά στην ιστορία τα αγαθά έχουν μετατραπεί σε οικονομικά ε, μέσα. Έχουμε... Αυτό έχει συμβαλεί σε δύο ε, παγκόσμιε επιστημιστικέ κρίσει τα τελευταία λίγα χρόνια. Δεν πρόκειται μόνο για θέμα κοινωνική δικαιοσύνη, αλλά και για θέμα γεωπολιτική σταθερότητας ε, στις χώρες, ε, στις στοχές χώρες με προβλήματα επισητιστικά. Δεν υπάρχει δυνατότητα στις χώρες όπου ο κόσμος ε, ξοδεύει 10% των εισοδημάτων του στο τρόφιμα οι συνέπειε φαίνονται αμελητέ. Ωστόσο, στι χώρε όπου αυτό το ποσοστό είναι το 70%, τα αποτελέσματα είναι καταστροφικά. Η πείνα προκύπτει από την ένδυα όταν οι τιμές των τροφών ψηλέ και όταν ε, οι άνθρωποι δεν μπορούν να καλύψουν τις βασικές, βασικές τους ανάγκες. Οι άνθρωποι το αντιμετωπίζουν αυτό ε, τρεφόμενοι λιγότερο, πουλώντας ε, περιουσία τους και χρεώνοντας την οικοκυριά τους. Αυτή η κατάσταση είναι εκτός ελέγχου και εφόσον δεν ληφθούν μέτρα κοινωνική προστασία, έχουμε να κάνουμε με ένα ζήτημα ζωή και θανάτου. Το γεγονό ότι ε, ο ανθρώπος ατόμων ε, που υφίστανται επισητιστική έλλειψη ε, έχει ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο είναι απαράδεκτο. Οφείλεται σε μεγάλο βαθμό σε μια φούσκα ουσιαστικά κερδοσκοπία που έχει περάσει τα τελευταία χρόνια και απαιτούνται μέτρα ώστε να αποφύγουμε μια άλλη μια κρίση επισητιστική. Σύμφωνα με τον ΦΑΟ, όλα τα γεωργικά αγαθά ήταν, ε, είναι σήμερα δύο φορές πιο ακριβά από ό,τι πριν από 10 χρόνια. Οι τιμές είναι 150% υψηλότερες από όταν το 2000. Υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία που υποστηρίζουν την ανάλυση ότι ένα μεγάλο κομμάτι αυτών των αυξήσεων τιμών σχετίζεται με την κερδοσκοπία. Θα ήθελα τώρα να επιστήσω την προσοχή σας στο γράφημα με τις ε, τιμές των τροφίμων που έχετε στο έγγραφο. 412 δισεκατομμύρια έφτασαν τα μέσα που βασίζονται σε αγαθά το Μάρτιο του 2011 αποτελούν ε, τεράστιο κομμάτι των συναλλαγών τουλάχιστον στις Ηνωμένε Πολιτείες η συμμετοχή τους διαστρεβλώνει τη λειτουργία της ε, αγοράς ε, και ο λόγος είναι ότι αυτές ορίζουν ε, τις τιμές σε ολόκληρο τον κόσμο. Διάφοροι εμπρογνώμονες υποστηρίζουν ότι η αύξηση των επενδυτών σε τέτοια παράγωγα έχει οδηγήσει σε αύξηση των τιμών και σε αστάθεια των τιμών. Η κερδοσκοπία σήμερα ήταν τόσο μεγάλη λόγω της ελευθέρωσης αγοράς τα τελευταία 10 χρόνια και θα συνεχίσει στην ίδια πορεία εκτός αν ληφθούν μέτρα για τον περιορισμό των ε, κερδοσκόπων στο ελάχιστο. Χρειάζεται να εισάγουμε κανόνες ε, που να διακρίνουν το hedging από την κερδοσκοπία και όχι απλά να κάνουμε τη διάκριση μεταξύ εμπορικών και οικονομικών φορέων. Τα ε, προϊόντα, τα οικονομικά προϊόντα που σχετίζονται με γεωργικά εμπορεύματα θα πρέπει να απαγορευτούν επειδή δημιουργούν τεχνητή ζήτηση. Ε, Σωστέ ρυθμίσεις για την πρόληψη των συστημικών κινδύνων είναι απαραίτητες και των πρακτικών χειραγώγηση χρειάζονται κανονισμοί ώστε να ε, αποκλειστούν ε, οι συναλλαγές επί εμπορευμάτων από, τις, από τα διάφορα κέντρα και τους τόπους διαπραγμάτευσης. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να περιοριστεί το μερίδιο του κάθε χειριστή σε κάθε αγορά. Επίσης θα πρέπει να βελτιωθεί η διαφάνεια στη θέση των συναλλαγών. Όλα τα παράγωγα που βασίζονται σε εμπορεύματα, τα παράγωγα επιμπορευμάτων θα πρέπει να ε, υπάρχουν μόνο σε ρυθμισμένες αγορές. Οι φορείς ε, ρύθμισης και εποπτείας θα πρέπει να ενισχυθούν ώστε να μην υπάρχει περίπτωση παράκαψης των απαγορεύσεων και των, και των ορίων. Επιπλέον, η χρήση απαγορεύσεων και ορίων δεν πρέπει να περιορίζεται στην άτακτη λειτουργία των αγορών στόχος του MIFID 2 θα πρέπει να είναι η πρόληψη και η εξάλληψη της υπερβολικής κερδοσκοπίας. Πιστεύουμε ότι το φαγητό αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα και προστατεύεται από την διεθνή διακήρυξη ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το να παίζει κανείς με αυτό είναι σαν να παίζει με τις ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων. Είναι το ίδιο σημαντικό όσο οποιοδήποτε άλλο περιουσιακό στοιχείο και δεν μπορεί να αφήνεται στις δύο των αγορών τα παράγωγα επιεμπορευμάτων και τα χρηματοοικονομικά παράγωγα δεν μπορούν να θεωρούνται ότι ανήκουν στην ίδια κατηγορία επενδύσεων. Πρέπει να ληφθεί προληπτική δράση για να διασωθούν οι ζωές. Έχουμε δημιουργήσει διάφορους μηχανισμούς αντιμετώπισης της αστάθειας των τιμών των τροφίμων, αλλά τίποτα που να μπορεί να, να αποτελεί προληπτικό μέτρο για αυτή την αστάθεια. Η κατάσταση λοιπόν είναι απαράδεκτη. Η συνθήκη της Λισαβόνας ε, έχει θέσει ως στόχους της Ένωσης την ε, μείωση της ε, φτώχειας και τη συνοχή για την ανάπτυξη. Αλλά σε τι μπορεί να χρησιμεύσει αυτή η ανάπτυξη και η πολιτική για την οποία εξοδεύονται 53 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο για να βοηθήσουμε τις ζωές των φτωχών στις αναπτυσσόμενες χώρες ενώ αφήνουμε τις χρηματαγορές να κερδοσκοπούν μαζικά στις βασικές επιστημικές ανάγκες των ίδιων ανθρώπων. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Ο κύριος Φέρπερ πρώτα έχει μια ερώτηση ως εισηγητής, έτσι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και ο τελευταίος γύρος, βέβαια, είναι πάρα πολύ σημαντικός Αναφέρθηκαν διάφορα ενδιαφέροντα θέματα. Ε, λίγες ερωτήσεις. Υπόθηκε από τον κύριο Τσερούτη ότι χρειάζεται ένας σαφής ορισμός των ε, παραγόγων των εξωχρηματιστηριακών παραγόγων, των OTC. Με το MIFIR λοιπόν με τον κανονισμό λαμβάνεται υπόψη και προσαρμόζεται σε ένα βαθμό και το ΕΜΙΡ. Ο ορισμός του ΕΜΙΡ είναι επαρκής ή όχι για σας. Γιατί δεν νομίζω ότι το μη φίτη, το ε, θα είχαν καθήκον να λύσουν κάποιο πρόβλημα το οποίο δεν έχει αντιμετωπίσει το ΕΜΙΡ. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ήταν αρκετά περίπλοκη ερώτηση. Και επίσης για τον κύριο Σλούτερ και την κυρία Ενρίκε. Κύριο Σλίτσερ ζητεί πλήρη εξαίρεση του δικού του τομέα και από τα position limits, αν τον κατάλαβα καλά. Για την κυρία Ενρίκ, μα λέτε ότι όχι χρηματοπιστωτικά παράγωγα ή πάντω όχι OTC στα τρόφιμα και αυστηρές, αυστηρά όρια στι στις θέσεις. Ε, ε, τώρα δηλαδή εμείς πρέπει να χωρίσουμε πολύ δύσκολες, ε, πολύ δύσκολες, ε, να αναλύσουμε άλλο πολύ δύσκολες εξισώσεις. Ανάλογα με τον τομέα θα πρέπει να το δούμε με το προϊόν. Ε, μήπως θα πρέπει να κοιτάξουμε μάλλον την διαφάνεια της αγοράς, δηλαδή τον χώρο της συναλλαγής περισσότερο, όπως είπε και η κυρία Ανρίκε, και εκεί να δώσουμε την έμφαση, ώστε να αντιμετωπίσουμε αυτές τις κερδοσκοπικές πιέσεις. Κυρίε μου, ότι συμφωνώ σε αυτό με την κυρία Ενρίκε για το, χρηματο... για το κερδοσκοπικό κομμάτι βέβαια, για το μερίδιο ε, της για θα πρέπει να το ε, χαλιναγωγήσουμε σε έναν βαθμό. Έχετε κάποια ιδέα για πιο συγκεκριμένε λύσεις. Γιατί η μία ακραία θέση είναι να μην γίνει, να μην πράξει κανένα έλεγχο, μια από την άλλη πλευρά ζητείτε να υπάρξει πάρα πολύ έλεγχο. Ναι, μήπως να ρωτήσουμε τον κύριο Τσερούτη, ο ίδιος τι πιστεύει. Ίσως να λύσει αυτό τη διαφορά ή την εξίσωση. Καλώ λέει ο κύριο Τσερούτη. Για να διευκρινίσω, γιατί ίσω να μην ήταν πολύ σαφή τα όσα είπα, η θέση μου για το MIFID δεν ήταν ε, να επαναπροδιοριστούν τα εξωχηματοστηριακά παράγωγα, αλλά να καταστήσουμε τον ορισμό που ήδη υφίσταται στο MIFID από το από την αιτιολογική σκέψη 3-2 να περάσει ο ορισμός στο ε, κόρπους του νομοθετήματος και να καταστεί έτσι δηλαδή υποχρεωτικός. Δεν ξέρω αν ήταν σαφή τα όσα σας είπα. Αλλά ας το ξαναδοκιμάσω, το από Και για το ΕΜΙΡ που αναφέρατε πιστεύουμε ότι ανεξαρτήτως του υποτμήματος της χρηματοπιστωτικής αγοράς που θα προσπαθήσουμε να επαναπροσδιορίσουμε θα πρέπει να δούμε τι αποσκοπούμε σε σχέση με τα έξω χρηματιστηριακά πράγματα. Δηλαδή, από την εμπειρία που έχουμε τα τελευταία χρόνια, η αδίποτε ασάφεια προς τα θα είναι εις βάρος και της αγοράς τις λειτουργίες τις αγορά λειτουργίες αγοράς και τελικά του κάθε ενός από τους παράγοντες που μετατέχουν σε αυτήν. Και εν μου επιτρέπετε, για τα όρια, για τα κοινοτικά όρια και τα, για τα κοινοτικά παράγωγα και τα όρια ως προς τις θέσεις, position limits, θα συμφωνήσω με τα όσα είπε η κυρία Ενρίκες, ότι είναι πολύ σοβαρό όλα αυτά τα θέματα κτλ. Δεν είναι όμως πουθενά δεδομένο ότι η λεγόμενη κερδοσκοπία προξενεί αυτή καθεαυτή την πτυτικότητα των τιμών. Αλλά και πάλι όπως είπα είναι δύσκολο το να κρίνει κανείς για τα τελευταία τέσσερα χρόνια έχουμε δει πολύ παράξενες εξελίξεις και ενοχλητικές. Ε, πάντως, πιο στοχευμένα μέσα ως προς τις θέσεις, τα όρια θέσεις, τα position limits και τους τελευταίους μήνες αυτών, των position limits, νομίζω μπορούν να φέρουν αποτέλεσμα ικανοποιητικό που θα καλύπτει και ε, κατ' επέκταση ή κατά προβολή καλύτερα ολόκληρο τον κύκλο της σύμβασης. Αυτό είναι καλύτερο νομίζω από το να προσπαθήσουμε να ξανασχεδιάσουμε ολόκληρη την αλυσίδα. Με συγχωρείτε, δεν... Ε, ε, έχουν ασκήσει αγωγή οι Ηνωμένε κατά του FTC για κάποιο ζήτημα σχετικό. Ναι, ξέρετε, δεν είμαι ειδικό στα θέματα των αγορών, ε, της αγοράς των Ηνωμένων Πολιτειών. Ναι, ούτε εγώ είμαι ειδικό, λέει ο κύριο Σλούτερ, αλλά θα προσπαθήσω, κύριε Φέρμπερ, να δώσω απάντηση στην ερώτησή σα. Μεταξύ της κυρίας Ενρίκες και των δικών μου δηλώσεων δεν βλέπω διαφορά εγώ τόσο μεγάλη. Γιατί είπε η κυρία Ενρίκες ότι πρέπει να γίνει διάκριση μεταξύ του χάτσιν και της κερδοσκοπίας. Αυτό λέμε κι εμείς. Εάν μιλούμε για πραγματική εξασφάλιση προθεσμίων, προθεσμιακών συμβάσεων δηλαδή, θα πρέπει αυτό να το δεχθούμε και ως δυνατότητα προστασίας της αγοράς της πώληση ε, πρώτων υλών ε, και προϊόντων. Για positions limit είμαι κατά και πάλι με παράδειγμα από το δικό μου τον κλάδο. Γιατί πώς λειτουργεί αυτό. Έρχεται μια αυτοκινητοβιομηχανία για να συστήσει μαζί μας την χρήση του ε, αλουμινίου, την αγορά δηλαδή αλουμινίου, χρήση καταρχάς στο δικό τον κλάδο και πρέπει στην περίοδο αυτή την ε, επταετή της παραγωγής του αυτοκινήτου που θα μπει στην αγορά στα τρία χρόνια να προβλέψουμε και την πτητικότητα του κινδύνου Άρα λοιπόν αν είχαμε position limit που ενδεχομένως θα έσχε για τρία χρόνια, ούτε και τον οδηγό, θα, τον ιδιοκτήτη δηλαδή, του αυτοκινήτου θα ε, εξυπηρετούσαμε, ούτε και εμάς, ούτε και κανέναν άλλον για να αποτρέψουμε ενδεχόμενους πιθανούς και πρόσθετους κινδύνους. Yeah, um, yes, just like to echo uh, what was... Ευχαριστώ. Θα ήθελα να αναφερθώ στην ε, ε, υπερβολική κερδοσκοπία ως προς τα limits που αποτελεί πρόβλημα γιατί παρεμβαίνει στη λειτουργία της αγοράς, διαταράσει την ενημέρωση για τις τιμές, προξενία συμμετρική ενημέρωση, παρεμποδίζει τη λειτουργία των συναλλαγών, ενισχύει την κινητικότητα των τιμών και γενικότερα δεν επιτρέπει να είναι ορατή η ε, κατάσταση που επικρατεί στις αγορές. Αυτό λοιπόν έχει κριθεί ήδη και η UNCTAD το 2009 έχει κρίνει ότι ε, επιδεινώνονται, επιδεινώνονται σε αγορές εξαιτίας αυτών των ε, ορίων. Και μάλιστα ακούστηκε ότι το New York Stock Exchange κάνει αγωγή κατά της CFTC ε, Πρόκειται δηλαδή για μια απόδειξη ότι μπορεί ο επενδυτής να παραβλαφθεί, να υποστεί σημαντική ζημιά λόγω αυτών των ορίων και προσπαθούν να το παρεμποδίσουν. Οι σκιώδες εισηγητές τώρα. Παρακαλώ. Ο κύριος Κέβελος. Ευχαριστώ. Ο κύριος Σλίτερ. Προσπαθεί εδώ να υπερασπιστεί την ε, αναγκαιότητα να παραμένουν αυτά τα μέσα στη διάθεση της πραγματικής οικονομίας. Αντιλαμβάνομαι ότι η πραγματική οικονομία χρειάζεται ενδεχομένως στο hedging για να αντιμετωπίσει κινδύνους. Έστω. Πλην όμως, αυτό δεν μπορεί να μας κάνει να παραλέψουμε το γεγονός ότι υπάρχει και η κερδοσκοπία Και δεν πρέπει να λησμονούμε ότι και ο κλάδος της παραγωγής θα πρέπει και φερρυπίν αποθηκευτικό χώρο να μισθώσει και διάφορα άλλα πράγματα. Εξαρτάται δηλαδή από πάρα πολλούς διαφορετικούς ε, Παρά πολλέ άλλε διαφορετικέ κατηγορίε τιμών που μπορεί να παρουσιάζουν επιτητικότητα και για τι οποίε δεν υπάρχει σχετική προστασία. Ω εκ τούτου, γιατί θέλετε εσεί ε, να προστατευτείτε σε σχέση με αυτό και με κάτι, με κάτι άλλο. Όλη αυτή η πτητικότητα υπάρχει και ρωτώ εάν θα έπρεπε να προσπαθήσουμε να την ε, ε, καταπολεμήσουμε και να εισαγάγουμε κανόνες διαφάνειας στην αγορά. Κύριε Σλίτσερ, το ότι δεν μπορώ εγώ να σχολιάσω τις επαγγελματικές πρακτικές τραπεζών, αλλά μια και είμαι 40 χρόνια σε αυτόν τον κλάδο των πρώτων υλών, θα πρέπει να σας διαβεβαιώσω ότι και από και πριν από 35 ακόμα χρόνια υπήρχαν τράπεζες οι οποίες ακολουθούσαν ε, τέτοιο πρότυπο χρηματοδότησης ε, στον χώρο των πρώτων υλών, δηλαδή χρηματοδοτούσαν και τους αποθηκευτικούς χώρους. Βέβαια αυτό έχει ενισχυθεί σε φαινόμενο υπερβολικά τα τελευταία χρόνια, το παραδέχομαι και ως εκ τούτου λέω ότι εφόσον πρόκειται για πραγματική αγορά, έστω και αν υπάρχει το φαινόμενο αυτό, πρέπει να παραμείνουμε εκτός από τη MIFID και επιμένω σε αυτές τις δηλώσει. Ευχαριστούμε κύριε Σούμπερ, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Δύο εντελώς ε, διαφορετικούς τομείς θέλω να θίξω, αναφερόμενοι στον κατάλογο που έχουμε. Η κυρία Ρώση ίσως να είναι πιο κατάλληλη να μου απαντήσει στην πρώτη μου ερώτηση. Έχει να με την κατηγορία των OTF, των Μηχανισμών Οργανωμένων Διαπραγματεύσεων, έτσι όπως εμφανίζονται στο κείμενο της Κομισιόν, και πώς θα είναι αρκετά ελαστικοί ώστε να καλύπτουν όχι μόνο τις πλατφόρμες διαπραγματεύσεων για τα παράγωγα, αλλά να χρησιμοποιούνται και για την ε, ρύθμιση. Από ό,τι καταλαβαίνω εγώ, εδώ υπάρχει ένα θέμα με τα Procrossing Networks έτσι όπως ορίζονται, γιατί οι επενδυτές χρησιμοποιούν την αρχή των Brooks και αυτό δεν θα γίνεται πια στα OTF. Οπότε οι επενδυτές δεν μπορούν να αναλάβουν κινδύνους αντισυμβαλόμενου. Αυτό το οποίο προτείνεται δηλαδή δεν είναι βιώσιμο. Οπότε, αν πρέπει να βασιστούμε στο μοντέλο της εσωτερήκευσης, τι αλλαγές πρέπει να γίνουν στο καθεστώς αυτό για να μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε καλύτερα, αντί για να έχουμε OTF. Και όσον αφορά τώρα τα παράγωγα επί εμπορευμάτων, αντιλαμβάνομαι και τις δύο πλευρές, αλλά ε, μία, ένας περιορισμός θέσης μπορεί να είναι κατάλληλος. Μήπως γίνεται κατάχρηση τελικά στις αγορές που το χρησιμοποιούν. Και μήπως τελικά πρέπει να υπάρξει ένα άλλο μέσο, πιο ίσως περίπλοκο, το οποίο επιτρέπει καλύτερη εποπτεία για την διαχείριση της θέσης και όχι καθορίζοντας μόνο κατόφλια, τα οποία όμως υπερβαίνονται. Κύριε Ρος, μείνατε εδώ παραπάνω και να που εξακολουθούν να σας έρχονται ερωτήσεις. Ναι, ακριβώς όπως είπατε έμεινε εδώ παραπάνω και να τώρα. Λοιπόν, είναι ένα ιδιαίτερα περίπλοκο ζήτημα αυτό. Ακόμα και ερώτηση νομίζω περιγράφει πόσο περίπλοκο είναι το ζήτημα και πόσο διαφορετικού τύπου διαπραγματεύσεις και διαδικασίες διαπραγματεύσεων και συστήματα διαπραγματεύσεων υπάρχουν που δεν είναι δυνατόν να ταξινομηθούν όλα και να μπουν σε έναν ενιαίο ορισμό. Δεν υπάρχει κάτι επίσημο. Αυτή είναι η θέση μου και είναι κάτι το οποίο κοιτάμε στις αναλύσεις ε, που κάνουμε για να δούμε πόσο διαφορετικά συστήματα διαπραγματεύσεων καλύπτονται μαζί. Οπότε, επιτρέψτε μου να το σκεφτώ και αργότερα να σας πω ποιες κατηγορίες, ποια συστήματα μάλλον θα μπορούσαν να ενοποιηθούν κάτω από μια κατηγορία. Ο Πρόεδρος, ευχαριστώ. Άλλη ερώτηση. Παρακαλώ, κύριος Κλούτε. Ευχαριστώ, Ζαν Πολ. Θα ήθελα να επισημάνω ή να παρατηρήσω, αν θέλετε, ότι τους τελευταίους μήνες στο γερμανικό τύπο ε, διεξάγεται ένας δημόσιος διάλογος ο οποίος έχει να κάνει με την κερδοσκοπία τόσο στο, θέμα, στο χώρο των τροφίμων όσο και στις πρώτες ύλε. Και εφόσον υπάρχει ο προβληματισμός πρέπει να δώσουμε μια απάντηση πολιτική, δεν μπορούμε να το αγνοήσουμε δηλαδή. Η κυρία Ενρίκες νομίζω ξεκάθαρα είπε ότι υπάρχουν ζητήματα δια, ε, διαφύλαξης προστασίας ε, της ε, επιβίωση του ανθρώπου, αλλά και ζητήματα δεοντολογικά, όχι μόνο οικονομικού ή πολιτικού χαρακτήρα. Και αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Ε, Επίση, βέβαια, διαπιστώνουμε από τη συζήτηση ότι είναι καθόλου εύκολο το να κρίνει κανεί ε, κατά τρόπο ισοδή και όλα αυτά τα πράγματα. Και γι' αυτό θα έλεγα πρώτα απ' όλα. Θα ρωτούσα για τον κύριο Σλούιτσερ αλλά και για την κυρία Ενρίκε. Εάν ενδεχομένως αντί να μιλούμε για position limits, να αποκλείουμε από τις ε, προθεσμιακές αγορές αγαθών την κερδοσκοπία, απλώς εδώ τους κερδοσκόπους. Νομίζω ότι υπάρχει κάτι τέτοιο ήδη στις Ηνωμένες Ή μη τι άλλο για την αγορά αργύρου από ό,τι είχα ακούσει πριν από ένα διάστημα τουλάχιστον. Η ίσχυη απαγόρευση τη κερδοσκοπία των κερδοσκόπων δεν μπορούσα να συμμετάσχει στην αγορά. Αλλά όπω είπε και ο κύριο Γκέμπελ, πώ μπορούμε να το ορίσουμε αυτό, πώ μπορούμε να περιγράψουμε αυτό τον κλάδο και να αποτρέψουμε καταστρατηγήσει ενδεχομένω τη ομοθοσίας αυτή, ώστε να παραμείνει η σταθερή αγορά. Το ένα είναι αυτό, το άλλο είναι η διαχείριση των ε, θέσεων, position management, που βλέπω, τουλάχιστον καταλαβαίνω από την δήλωση της Επιτροπής, ότι είναι πιο ασθενής, ασθενές μέσων από το position limits, από τα όρια στις θέσεις. Πώς το βλέπετε σε αυτό ως ειδική. Τρίτη και τελευταία ερώτηση ίσως για τον κύριο Τσερούτη περισσότερο. Υπάρχει μια ειδική εποπτική αρχή για το εμπόριο σε τρόφιμα, συναλλαγές σε τρόφιμα και πρώτες ύλες. Μήπως θα έπρεπε να ρωτήσουμε και εμείς ε, να διερευνήσουμε τη δυνατότητα να εισαχθεί μια αντίστοιχη αρχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι ως τέταρτη εποπτική αρχή, αλλά με μια άλλη εναλλακτική φερρυπίν στο πλαίσιο της ΕΚΑ ή σε ένα ιδιαίτερο στην ιδιαίτερη διεύθυνση της ΕΚΑ, μια μονάδα η οποία θα ασχολείται ειδικά με το θέμα αυτό. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Πριν, το δώσω το λόγο για να απαντήσουν οι προσκεκλημένοι μας, ο εισηγητής παρακαλώ. Ναι, ευχαριστώ. Μια και είναι και οι δύο κυρίες από το δεύτερο πάνελ ακόμη εδώ, θα εκμεταλλευτώ και εγώ την παρουσία τους. Είπατε κυρία Ανρίκες, κύριε Σλούιτερ, ότι ναι μεν υπάρχει ένα, μια αγορά αγαθών και είπατε ότι θέλετε να αφήσετε αυτή την αγορά ελεύθερη να δρά σε σχέση με τις τράπεζες, αλλά όταν έρχεται η ώρα οι τράπεζες να παρέμβουν στην αγορά αυτή, τότε πρέπει να την προφυλάξετε. Να την προφυλάξουμε εμείς. Είναι δυνατόν να έχουμε και την πίτα ολόκληρη και τον σκύλο χορτάτο. Και εμεί ω ρυθμιστική, η ρυθμιστική αρχή, εν περιπτώσει, πώς μπορεί να παρεύει σε, αυτή, την, ε, σε αυτό το πεδίο. Και πώς θα κρίνει αν πρόκειται για μια ε, απλή συναλλαγή ή αν πρόκειται για προϊόν κερδοσκοπία. Ο οι, παρέχοντες στην υπηρεσία μπορούν να δουν μια τέτοια διάκριση. Ευχαριστούμε. Να ξεκινήσουμε με τη σειρά. Να απαντήσετε ίσως, κυρία Ρίκες, πρώτα στην ερώτηση του κύριου Κλούτια και του εισηγητή. Έτσι, γιατί και σε εσά απευθύνθηκε κάποια ερώτηση. Ναι, λέει κυρία Ρίκη. θα προσπαθήσω να απαντήσω στις διάφορες ερωτήσεις. Μια από τις κριτικές που ακούμε για την MIFID είναι ότι δεν εφαρμόζεται ρυθμισμένα και αυτό είναι που μειώνει τους ελέγχους και αφήνει περιθώρια για καταχρήσεις. Επίσης υπάρχουν κάποιοι όροι οι οποίοι δεν ορίζονται σαφώς και συγκεκριμένα. Βέβαια υπάρχουν κάποιες εναλλακτικέ ε, λύσεις που προτείνονται αλλά πάλι παραμένει μεγάλο περιθώριο ερμηνείας. Η γνώμη μου είναι ότι πρέπει να προσπαθούμε να είμαστε όσο μπορούμε πιο συγκεκριμένοι και να ορίζουμε τα κριτήριά μας και τις παραμέτρους μας όσον αφορά την κερδοσκοπία και για τους ε, οικονομικούς συμβολόμενους και για τους μη οικονομικούς. Τώρα, ποια είναι τα πλονεκτήματα Τη αγορά παραγόγων επί εμπορευμάτων και ποια είναι η σφορά του στην πραγματική οικονομία και κατά πόσο ε, συνοδεύονται τα πλεονεκτήματα από κινδύνους. Κοιτάξτε, ε, η κερδοσκοπία δεν είναι επένδυση. Άλλο οι εμπορικοί παράγοντες, άλλα τα άλλοι hedgers, δηλαδή τα κεφάλαια κινδύνου και άλλο η κερδοσκοπία αυτή καθεαυτή. Πρέπει να κάνουμε διάκριση ανάμεσα αυτά. Ο κύριος Λούτα. Ευχαριστώ. Πολύ ευχαριστώ. συμφωνήσω με την προλαλή σας. επί της αρχής συμφωνούμε βεβαίως. 100% και πιστεύουμε ότι οτιδήποτε δεν μπορεί να αποτελέσει ικανοποίηση υλική ανάγκης μπορεί να μπει στον τομέα της κερδοσκοπίας και όλα τα υπόλοιπα ανέκουν στην πραγματική οικονομία. Για τα position limits, στον τομέα τουλάχιστον των πρώτων υλών, τα βλέπουμε διότι ο, η ποσότητα μιας παραγόμενης πρώτης ύλης είναι ως εκ περιορισμένη δεν μπορούμε να έχουμε ελεύθερα position limits. Είπα και νωρίτερα ότι όλα αυτά έχουν εφαρμογή στην πραγματική οικονομία και άρα θα πρέπει να αντιστοιχούν και στην πραγματική οικονομία. Ναι και συμφωνούμε όλοι το θέμα είναι ανησυχητικό. Πολλά ζητήματα τίθενται και από κοινωνική άποψη. Δεν αποτελεί μόνο ζήτημα η αποτελεσματική λειτουργία της αγοράς αλλά και το κατά πόσο υπάρχει ακαιρεότητα από κοινωνική άποψη. Χωρίς να μακρηγορήσω, υπάρχει κοινωνική αξία όσον αφορά τη χρηματοοικονομική συμμετοχή σε μια συνεκτική αγορά. Το θέμα να βρούμε την ισορροπία μεταξύ της υπερβολικής κερδοσκοπίας και αυτής της κοινωνικής αξίας. Έχουμε πολλά παραδείγματα αυτής της κοινωνικής αξίας. Μην δαιμονοποιούμε λοιπόν όλη τη συμμετοχή σε χρηματοοικονομικές αγορές. Έχουν υπάρξει πολλά ωφέλη, επίσης αναγνωρίζουμε ότι υπάρχει μια μυστηριώδης ε, σχέση μεταξύ της υπερβολικής ε, χρηματιστικοποίησης κατά κάποιο τρόπο των εμπορευμάτων και της ε, αστάθειας έγιναν συζητήσεις και υπάρχει μια εκθέση της Κομισιόν από τον τελευταίο Φεβρουάριο για να προσδιοριστεί κατά πόσο υπάρχει αυτός ο συσχετισμός. Εγώ δεν έχω διαποδεικτικά στοιχεία, αλλά ωστόσο έχει ενδιαφέρον ε, και αφορά τα κοινωνικά ζητήματα. Τώρα, όσον αφορά την ερώτηση που μου τέθηκε, πιστεύω ότι η δυσκολία είναι να βρούμε τη σωστή ισορροπία μεταξύ της μη ε, εξάλληψης ουσιαστικά της κοινωνικής αξίας τη συμμετοχή ε, στην αγορά και της αποφυγής της ε, κερδοσκοπίας και της αστάθειας των τιμών. Εδώ στην πρώτη της Επιτροπής αναφέρεται position limit ή εναλλακτικές διευθετήσεις. Η παροχή όριων μπορεί να είναι πολύ αποτελεσματική να επιτύχει αυτούς τους στόχους αυτό ήταν ουσιαστικά αυτό που θέλαμε να πούμε. Τέλος, ε, δεν είμαι σίγουρος κατά πόσο χρειαζόμαστε μια άλλη αρχή για αυτό το ζήτημα. Ωστόσο, σε τέτοια περίπτωση, εμείς ε, είμαστε υπέρ. Βρισκόμαστε σε ένα υψηλά ρυθμισμένο περιβάλλον σε όλες τις αγορές. Έχουμε συνεργαστεί με τις ρυθμιστικές αρχές. Οτιδήποτε θα μπορούσε να βελτιώσει τον τρόπο λειτουργίας των αγορών και την κοινωνική του ωφέλεια θα ήταν ευπρόσδεκτο από εμάς. tu as été visé par Marcus. C'est les vieux souvenirs du mandat Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εκμεταλλεύομαι την ευκαιρία για να πω μερικά λόγια σε αυτή τη συζήτηση. Θα πάω λίγο πιο πίσω στη συζήτηση. Έγινε μια συζήτηση για το τι πρέπει η ευρωπαϊκή η κεφαλαία αγορά να εξυπηρετεί πραγματικά, ποιοι είναι οι, οι δικαιούχοι ουσιαστικά των ωφελών όλων αυτών των ρυθμίσεων, ποιος είναι ο δικός τους ρόλος. Έχοντας αυτό το ρεύμα νέων ε, ρυθμίσεων στην Ευρώπη, σημαίνει ότι όλο και περισσότερες ε, οικονομικές εταιρείες μετατρέπονται σε χρηματοοικονομικές εταιρείες λόγω των διαφορών κανονισμών απαγόρευσης των χρηματοοικονομικών ρυθμίσεων. Έχουμε ειδικά μεγάλες εταιρείες που ουσιαστικά αυτοχρηματοδοτούνται. Το κάνουν από τις αγορές, ε, απευθείας από τις κεφαλαίες αγορές. Κινούμαστε λοιπόν προς αυτόν τον αμερικανικό τρόπο χρηματοδότησης των πραγματικών οικονομικών μας αναγκών. Αυτό σημαίνει ότι και σε αυτή τη συζήτηση για το ποιο ουσιαστικά πραγματοποιεί πραγματικές συναλλαγές και ποιος είναι ο τελικός, ο απότερος στόχος όλων αυτών, εδώ η εικόνα είναι λιγάκι πιο θολή θα πρέπει να φροντίσουμε να έχουμε ίσους κανόνες ανταγωνισμού για τις επενδυτικές εταιρείες και τις πραγματικές οικονομικές εταιρείες όταν αυτές κερδοσκοπούν εντός εισαγωγικών ή πραγματοποιούν συναλλαγές στην αγορά. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο έχουμε συζητήσει στην ομάδα Business Europe και μέχρι στιγμής δεν έχουμε καταφέρει να βρούμε αυτόν τον ορισμό που ζητάει ο εισηγητής τι είναι κερδοσκοπικό και τι δεν είναι. Φυσικά οι χρηματομεζίτε θα αξιοποιήσουν την ευκαιρία σε περίπτωση που αυτός ο ορισμό δεν είναι σαφή. Πιστεύω λοιπόν ότι όλη αυτή η συζήτηση του να προσπαθούμε να μπούμε στο μυαλό κάποιου είναι εξαιρετικά δύσκολη. Και φυσικά αυτή η τάση προς πιο προς εταιρείε ε, που χρηματοδοτούνται με αμερικανικό τρόπο. Θα πρέπει επίσης να βρεθεί ε, στο επίκεντρο των συζητήσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ κύριε Ρος. Ε, νομίζω ότι σας τα σας μια ερώτηση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρέπει να πω ότι συμφωνώ απόλυτα με ορισμένους από τους προλαλήσαντες το να προσπαθούμε να καθορίσουμε τι είναι hedging και τι είναι κερδοσκοπία είναι εξαιρετικά δύσκολο. Είναι δύσκολο να καθοριστεί ο στόχος, ο σκοπός της συναλλαγής ε, ακόμη και ως χρηματοοικονομική εταιρεία όπως είστε εσείς ε, και στις συναλλαγές επί εμπορευμάτων θα δυσκολευτεί το, η δραστηριότητά σας από ορισμένε ε, πτυχές. Είναι δύσκολο να καθοριστεί τι είναι hedging και τι είναι κερδοσκοπία. Τα όρια είναι πολύ δύσκολο να χαραχθούν. Πιστεύω ωστόσο ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε να κάνουμε άλλη μια προσπάθεια γι' αυτό. Ευχαριστώ. Υπάρχουν άλλες ερωτήσεις από τους συναδέλφους. alors je vais donner δεν βλέπω να υπάρχουν άλλε ερωτήσεις. Θα δώσω το λόγο λοιπόν στον κύριο Σιγητή ώστε να μας δώσει τα συμπεράσματα από αυτήν την ακρόαση. Ευχαριστώ πολύ όλους τους ομιλητές για την παρουσία τους και τις ομιλίες τους οι οποίες μας διαφώτισαν για ένα πολύπλοκο θέμα το οποίο ίσως να μην είναι ιδιαίτερα δημοφιλές αλλά που σίγουρα συνεπάγεται πολλή εργασία για εσάς. Πρόεδρε, ευχαριστώ και εγώ βεβαίως θα συμφωνήσω και θα ευχαριστήσω από πλευρά μου τους ε, παρεμβαίνοντας από τα τρία πάνελ. Ε, Ιδιαίτερος δε, διότι μας άφησαν τόσα πολλά ερωτηματικά χωρίς απάντηση. Στα οποία θα πρέπει να δώσουμε εμείς απαντήσεις ως νομοθέτες. Είναι το καθήκον μας άλλωστε αυτό σε ένα τομέα στον οποίο επικρατεί η ασάφεια να δώσουμε απαντήσεις και ασφάλεια δικαίου. Και Βεβαίω, δεν μπορέσαμε να, δώσουμε, να συστήσουμε κάθε λεπτομέρεια τη πρόταση ΜΕΦΙΝΤ, αλλά πάντω τα κύρια ζητήματα, τα πολιτικά ζητήματα, πιστεύω μπορέσαμε να τα δούμε στη διάρκεια αυτή τη ακρόαση. Πολύ υλικό για σκέψη δόθηκε, θα το λάβουμε υπόψη ασφαλώ. Και επισημαίνω ότι έχουμε επεξεργαστεί ένα ερωτηματολόγιο Διαπιστώνω δεν μετά καταπλήξω ότι η Financial Watch μας ε, προεξήγγειλε τροπολογίες. Είπε ότι θα καταθέσει προτάσεις ε, για τροπολογίες στα κείμενά μας. Εν πάση περιπτώσει γιατί όχι, για λόγους διαφάνειας, πολύ ευχαριστώ να δούμε ό,τι πρόταση έχει. Ας χρησιμοποιήσει το ερωτηματολόγιο και νομίζω ότι είναι αρκετά λεπτομερές ε, και διεξοδικό πολύ περισσότερο από ότι αυτό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επίσης, τελευταία ανάλυση έχουμε πολύ πιο στοχευμένη προσέγγιση σε σχέση με την Επιτροπή, η οποία έπρεπε, αφού ξεκινούσε τη δουλειά, να κάνει μια πιο γενική ε, προσέγγιση. Εν πάση περιπτώσει, εάν έχω ορθή ενημέρωση από τη Γραμματεία, προβλέπεται να συζητηθεί για πρώτη φορά στις 13 Φεβρουαρίου ε, η έκθεση. Άρα ένα μήνα μετά τη λήξη προθεσμίας για την κατάθεση παρατηρήσεων στο ερωτηματολόγιο, η απαντήσεων στο ερωτηματολόγιο. Άρα έχουμε ένα μήνα στη θέση μας ανάμεσα στο ερωτηματολόγιο και στην έκθεση με συνεδρίαση στο Στρασβούργο σημειώνω Δευτέρα βράδυ, άρα με εγγύηση μεγάλης προσέλευσης αφού θα είναι στο Στρασβούργο. Ευχαριστώ τους συναδέλφους, προσβλέπω στην περαιτέρω συνεργασία και είμαι βέβαιος ότι η επόμενη χρονιά θα σημάνει πολύ στενή συνεργασία μεταξύ μας. Η διαδικασία δεν είναι εύκολη. Έχουμε ε, θέματα, τομείς, στους οποίους πρέπει να δώσουμε απαντήσεις όχι μόνο τεχνικές, αλλά και πολιτικές. Και αυτή είναι η δουλειά μας, τελευταία ανάλυση. Και κάπου στα μέσα του 2012 θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε το Συμβούλιο με την διαπραγμάτευση για τις διαφορετικές μας θέσεις και φαντάζομαι το δεύτερο εξάμεινο του 2012 θα είναι μάλλον συναρπαστικό χρηματοπιστωτικό πλαίσιο, νομοθετικά κείμενα δηλαδή το χρηματοπιστωτικό και ε, πλαίσιο και ε, μικρό πράγματα ψίχουλα όπως το MIFID θα μας απασχολήσει το δεύτερο εξάμεινο του 2012. Άρα φαντάζομαι ότι θα έχουμε πολλή δουλειά. Καλό λοιπόν τους συναδέλφους να συνεργαστούμε όλοι μαζί για να έχουμε στον δυνατόν καλύτερη λύση, μία λύση, μία πρόταση, η οποία θα δώσει σωστέ απαντήσει στη ρύθμιση των χρηματοπιστωτικών αγορών. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρο. Ευχαριστώ όλου όσοι έλαβαν τον λόγο σήμερα, όλου του συναδέλφου. Και μια και έχουμε αρκετό κόσμο μέσα στην αίθουσα, επιτρέψτε μου να επισημάνω ότι το 2011 η Οικονομική και Νομισματική Επιτροπή μα, που έχει πάρα πολύ μεγάλο φόρτο εργασία, διεξήγαγε 48% περισσότερες συνεδριάσεις από το προηγούμενο το 2010 δηλαδή. Πράγμα το οποίο αποδεικνύει ότι το Κοινοβούλιο δουλεύει πολύ σκληρά. Προσεχή συνεδριασή μας στις 12 Δεκεμβρίου και επί τη ευκαιρία θα έχουμε και την ακρόαση του υποψηφίου για το διευθυντικό όργανο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ευχαριστώ πολύ. Πέρα στη συνεδρία σας.